Buenos días. Καλή σας ημέρα. Ο κ. Κρίστεσεν δεν έχει κάρτα ψηφοφορίας, οι υπόλοιποι ας τις δοκιμάσουν. Ε, τον κύριο Κρίστεσεν θα τον καταμετρούμε χωριστά. Κανείς άλλος? Ωραία. Σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μια μικρή τροποποίηση στην αρχή των ψηφοφοριών θα θέσουμε σε ψηφοφορία την έκθεση Ρωμέβα για τα παραλίευματα ειδών. Είναι ε, πρόορη δεύτερη ανάγνωση. Τίποτα άλλο. Ο κ. Πρεσέδο μου είπε ότι θα φτάσει καθυστερημένα και μου ζήτησε να μετακινήσουμε το θέμα του. Του είπα όμως ότι δεν είναι δυνατόν διότι έχουμε εκθέσεις. Οπότε σας ζητάει να τον συγχωρήσετε που θα λείπει. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσει του Προέδρου δεν έχουμε τίποτα. Ο κ. Ρωμέβα είναι εδώ. Ας περιμένουμε τον κύριο Μέβα να καθίσει. Ελπίζω να μην χάσουμε ψηφοφορία για μία μόνο ψήφο. Περνάμε στην ψηφοφορία... Συγγνώμη. Ναι. Τη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης κύριου Ρωμεβά. Ξεκινάμε. Ya, ya, bueno. Cerramos. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Πολιετές πρόγραμμα ανασύστασης ε, του, ε, ε, στρουτών του, Ατλαντικού, του Ανατολικού Ατλαντικού, έκθεση του κυρίου Ρωμέβα. Δεν δουλεύει το μηχάνημά σας. Δεν είναι ανοιχτή η ψηφοφορία, οπότε μην προσπαθείτε να ψηφίσετε. Ωραία. Για να δούμε αν λειτουργεί. Είμαστε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Πολιορχητέ σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Τροπολογία υπαριθμών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λειτουργούν όλα. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ξεκινάμε. Λήξη πληροφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4. Έναρξη πληροφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Ε, ψηφίζουμε την πρόταση του σύνολό τη. Έναρξη πληροφορία. Λήξη εγκρίνεται. Και το νομοθετικό ψήφισμα έναρξη ψηφοφορίας, λήξη πληροφορία εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Ρωμέβα. Περνάμε στην έκθεση για την κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του Ευρωπαϊκού Τομέα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ταϊλάνδη. Καταρχήν ψηφίζουμε την ε, συμβαστική πρόταση παρθμών 1. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση παριθμών 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση παριθμών 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Είναι τα 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Ε, έναρξη ψηφοφορία, συγγνώμη. Λέξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Τη κυρία Πατράου. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Συμβασμό 5. Έναρξη. Λεξή. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Έναρξη. Λεξή. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ίντα 1 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ίντα 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός παριθμών 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός παριθμών 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Όχι. Α, απορρίπτεται. 8-8. Για την τροπολογία 6 μιλάμε. Τροπολογία 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 9. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Η 8 έτσι. Ωραία. Τροπολογία 9. Έναρξη. Λήξη. Η 9. Την 9 ψηφίζουμε. Α, την 9, η 9 απορρίφθηκε. Η απορρίφθηκε, η 9 απορρίφθηκε. Με περνάμε στη οσφορία της τροποποιημένης έκθεσης. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές. Ευχαριστούμε. Περάμε στο επόμενο θέμα. Προ... Όχι έκθεση. Σημείο 6 πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δημοκρατία των Σεχελών. Όπω ξέρετε, τον Γενάρη κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το ζήτημα. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο ανα, ε, σύστασης της εισηγήτρας κυρίας ε, Πατράου Νέβες, στην οποία δίνω και το λόγο. Κυρία Πατράου, Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων σας υπογράμμισα το ότι αυτή η πρόταση ε, συμφωνίας με τις Χέλες είναι πολύ ισορροπημένη, λογική και μάλιστα συμφέρουσα και για τα δύο μέρη. Τα μέλη που είναι εδώ σήμερα ήταν παρόντα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, οπότε θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω πολλά πράγματα. Άλλωστε, στην τελευταία μας συνεδρίαση είχα ήδη δώσει την εκθεσή μου προς μετάφραση Οπότε τη διαβάσατε αργότερα εσείς, τα είχα όμως πει και προφορικά. Σήμερα θα υπογραμμίσω τις πιο σημαντικές ε, πτυχές έκθεσής μου και ιδιαίτερα αυτές ε, τις οποίες ε, ανέπτυξα μετά την τελευταία μας συνάντηση. Και θέλω να σας αποδείξω ότι αυτή η έκθεση είναι ισορροπημένη, είναι καλύτερη από την προηγούμενη και κατά την άποψή μου θα πρέπει να εγκριθεί. Ο αληφτικός τομέας ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις Σεϊχέλες. Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία ο τουρισμός ήταν ε, ο κλάδος που είχε το μεγαλύτερο βάρος ε, στο ΑΕΠ των Σεϊχελών, όμως πλέον η αλία τον έχει ξεπεράσει. η αλία είναι πλέον ο κλάδος ε, που βαρύνει περισσότερο στην οικονομία των Σίχελων. Αντιπροσωπεύει το 31,4% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, ε, προ, προϊόντος. Συγγνώμη. Οι θέσεις απασχόλησης, έμεσες και άμεσες, που συνδέονται με την αλία είναι περίπου 5.000 κάτι που αντιπροσωπεύει το 10% του ε, ε, εργατικού δυναμικού της ε, επίσημης απασχόλησης στη χώρα. Είναι λοιπόν σημαντικός ο κλάδος αυτός. Γι' αυτόν τον λόγο και οι Σεϊχέλες ασχολούνται πολύ με αυτή τη συμφωνία, της ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επίση, είχα σχολιάσει και στην προηγούμενη συνεδρίασή μα το θέμα τη πειρατεία. Ο κίνδυνος αυτός όμως μειώνεται όσο περνάει ο χρόνος. Και η μείωση του ενδιαφέροντος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχει πλέον εξαφανιστεί ακριβώς διότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος πειρατείας. Ε, πλέον ε, ο αλληλευτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρεται και πάλι να αλλιεύει τα ύδατα των Σεχελών. Πρόκειται για αλλία των οειδών κυρίως κάποια, ένα μικρό αριθμό μεταναστευτικών ειδών. Κυρίως ε, ερυθρό τόνο του βορρά, κυτρινόπτερο τόνο και μεγαλόφθαλμο τόνο. Πρόκειται για είδη ε, τα οποία τυχαίνουν πλήρης ε, εκμετάλλευσης Ε, μάλιστα ο ερθρός τόνος είναι υπό εκμεταλλευόμενος αυτή τη στιγμή. Τα κράτη-μέλη τα οποία περισσότερο λειτουργούσαν και αλίευαν σε αυτά τα ύδατα, ε, ιδιαίτερα τα γαλλικά και ισπανικά γρηγρή, ε, είναι, είναι ιδιαίτερα τα ισπανικά και γαλλικά γρηγρή, ε, αλλά και παραγαδιάρικα, ε, τα οποία κυρίως είναι από τις Αιχέλες και τις ε, Φιλιππίνες, ε, λιγότερο δηλαδή ευρωπαϊκά σκάφη και περισσότερο ντόπια. Τα ευρωπαϊκά παραγαδιάρικα τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλείψει τη ζώνη αυτή. Αυτό το φαινόμενο ε, απηχείται και, στα, στον όγκο των αλλιευμάτων. Ε, έχουμε μείωση ε, από 48 σε 40 τον γρηγρή, από 12 σε 6 για τα παραγαδιάρικα. 14 συνολικά σκάφη λιγότερα λοιπόν από πλευρά του Ευρωπαϊκού ε, Στόλου ε, σε αυτό το καινούριο πρωτόκολλο σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό απηχεί το φαινόμενο της, ε, του μικρότερου ενδιαφέροντος από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον μας εξακολουθεί να υπάρχει το, το, τα σκάφη που έλειβαν τα τελευταία χρόνια ήταν ακόμα λιγότερα. Τώρα σε ό,τι αφορά το αντιστάθμισμα, η χρηματική αντιπαροχή, ε, και πάλι είναι λογική, στο προηγούμενο πρωτόκολλο είχαμε 16 περίπου εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, τώρα έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου για έξι χρόνια. Οπότε και η αντιπαροχή είναι απόλυτα λογική. Υπάρχει επίσης αύξηση της ε, υποστήριξης του κλάδου. Είναι σημαντικό αυτό και για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Αιχέλες. Σε ό,τι αφορά τις αλληλευτικές ε, άδειες, βλέπουμε μια αύξηση σε ό,τι αφορά τις ε, αξίες, τις, ε, το, το τέλος που χρειάζεται να πληρωθεί. Ε, συγκρίνουμε ένα πρωτόκολλο τριών ετών το προηγούμενο με ένα καινούριο πρωτόκολλο έξι ετών που είναι το καινούριο. Οπότε θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Το γεγονό ότι είναι εξαετέ το καινούριο πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα συμφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί προσφέρει μια σταθερότητα και περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού των αλληλευτικών δραστηριοτήτων στους επαγγελματίες αλληλείς. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι περνάμε από ένα πρωτόκολλο τριετούς διάρκειας σε ένα πρωτόκολλο εξαετούς διάρκειας. Να πω και δύο λόγια πρόσθετα σε σχέση με ό,τι είχα πει την, στην προηγούμενη μας συνάντηση. Από τότε ε, έχουμε πλέον την έκθεση για τον προπολογισμό της ε, Κομισιόν που υποστηρίζει ε, την ανανέωση της αλληλευτικής σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σεϊχελών. Η Επιτροπή Προπολογισμών λοιπόν μας στηρίζει Και επίσης να σας πω ότι ε, ήρθα σε επαφή και με την ε, πρέσβυρα των Σεϊχελών καθώς επίσης και τον πρόεδρο της ε, αλληλευτικής αρχής των Σεϊχελών. Συζητήσαμε τους όρους της συμφωνίας και μου είπαν και οι δύο και η πρέσβυρα και ο πρόεδρος ότι βλέπουν πολύ θετικά την έκθεση αυτή, την συμφωνία αυτή και οι ίδιοι θεωρούν ότι η συμφωνία είναι προς συμφέρον και των δύο πλευρών, πολύ ισορροπημένη. Εκτιμούν ιδιαίτερα την διαφάνεια και ενημέρωσαν επίσης ότι και ο κόσμος της Εχέλες βλέπει πολύ θετικά τη συμφωνία αυτή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ε, πολύ ορατή δεδομένου ότι υποστηρίζει και την στηρίζει μάλλον ε, οικονομικά και την κατάρτιση των αλλιών και την ε, δημιουργία υποδομών. Από την κοινή γνώμη διάκειται πολύ θετικά. Και ό,τι αφορά τι υποδομές, ε, τι λιμενικές υποδομές και τα λιμενικά έργα, για παράδειγμα, ε, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε την ε, καλύτερη επεξεργασία και μεταποίηση των αλλιευμάτων, την αποθηκευσή τους, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση, εμπορική εκμετάλλευση άλλων ειδών, τα οποία δεν εκμεταλλευόντουσαν στο παρελθόν. Δηλαδή βελτιώθηκε η διαφοροποίηση. Ε, επίσης αξιοποιήθηκαν ε, ε, μάλλον αυτά τα καινούργια είδη έδωσαν και καινούργιο εισόδημα. Σε ό,τι διάφορα τις υποδομές δημιουργήθηκαν καταφύγια για την μικρή κλίμακος Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στη μικρή κλίμακα και τη βιομηχανική αλεία. Γιατί έχουν, έχουν διαχωριστεί οι αλληλευτικέ ζώνε. Δεν συγκρούνται λοιπόν αυτέ οι δύο μορφέ αλεία. Και οι δύο αισθάνονται ότι καλύπτονται από αυτή την συμφωνία διότι βλέπουν και νιώθουν τα, τα ωφέλη που προκύπτουν. Επίσης μου είπαν η πρέσβηρα και ο πρόεδρος ότι είναι σημαντική η υποχρέωση χρησιμοποίησης τόπιων πληρωμάτων. Αυτό δεν είναι ότι προσθέτει τόσο πολύ στην απασχόλησή τους όσο στην κατάρτισή τους. το ότι δουλεύουν σε ευρωπαϊκά λευτικά σκάφη τους επιτρέπει να βελτιώσουν την κατάρτισή του τις γνώσεις τους και αυτό θα τους εξασφαλίσει αυτονομία στο μέλλον. Επίσης μου υποδείχθηκε ότι είναι σημαντική η επιστημονική έρευνα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και με το νέο πρωτόκολλο, ε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, άλματα θα έλεγα, στην ε, δημιουργία ενός ε, ε, Μια ομάδας ερευνητών, ντόπιων ερευνητών, που θα στηρίξει στο μέλλον τη διαχείριση του αλευτικού τομέα. Πολύ θετική λοιπόν η αντιμετώπιση της ε, συμφωνίας αυτής και από πλευράς ε, των ηγετών, των κυβερνώντων, όσο και από πλευράς του κόσμου της κοινής νόμης. Όλα τα στοιχεία λοιπόν μας οδηγούν στο να συμπεράνουμε ότι είναι μια ε, συμφέρουσα συμφωνία για όλους. Είναι μια συμφωνία καλύτερη από την προηγούμενη, κυρίως γιατί περνάμε από μια διάρκεια τριετή σε μια διάρκεια εξαετή. Αυτό το υποστηρίζουν όλοι οι δείκτες, όλα τα επιχείρηματα που οποία σας ανέφερα. Συνεπώς ε, ελπίζω ότι την ίδια γνώμη θα συμμεριστείτε και εσείς οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ για αυτή την εκτεταμένη παρουσίαση. πολύ δουλειά είναι σαφές ότι κάνατε. Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Μαρία Πατραονέβες για την εξαιρετική της έκθεση και την παρουσίαση της Συμφωνίας Αλληλευτικής Σύμπραξης με τις Σεϊχέλες. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω προς την Κομισιόν κυρίως. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχουν ξεχωριστές ποσοστώσεις για τους καρχαρίες ε, καθώς ε, και για τους ξηφίες και υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια παρεπίπτοντα αλλιεύματα, ωστόσο λέει ότι έχουμε έξι γρηγροί και περίπου το 30% είναι παρεπίπτοντα αλλιεύματα τέτοιων ψαριών στα μη ευρωπαϊκά σκάφη και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για τα ευρωπαϊκά σκάφη. Και αναρωτιέμαι επίσης τι ισχύει όσον αφορά τα φάτς, τις διατάξεις συγκέντρωσης εχθείων. Ποια είναι τα παρεπίπτωτα αλλιεύματα σε αυτή την αλία. Υπάρχει κάποιος περιορισμός ε, στη συμφωνία αυτή όσον αφορά τον αριθμό των διατάξεων συγκέντρωσης ισχύων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει κάποιο σχέδιο διαχείρισης αυτών των φαντ. Και τέλος, όσον αφορά την τομεακή βοήθεια. Βλέπουμε μικρή αύξηση. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιηθεί και η τελευταία ερώτηση είναι γιατί έχουν μειωθεί οι πληρωμές για τα αγριγρή τόσο πολύ. Έχουν μειωθεί σε περίπου 38 με 52.000 ε, το χρόνο για τα αγριγρή. Πώς, γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί έχει μειωθεί η τιμή αυτή. ενώ γενικά πληρώνουμε περισσότερο για τα λιεύματα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. thank you very much for... Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω ε, σκιώδη ε, των φιλελεύθερων θέλω να πω δύο λόγια. Εγώ ήμουν σε αντιπροσωπεία που πήγε σε Ιχέλες και έχω αυτό πλεονέκτημα. Εντυπωσιάστηκα πρέπει να πω από την συνολική κατάσταση εκεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη βιώσιμη ε, αλία και από την έκθεση είδα ότι για το μεγαλόθωμο και τον κυτρινοπό τόνο θα πρέπει να προσέξουμε να μην ξεπεράσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Να μην υπερ... Ε, εκμεταλλευόμαστε αυτά τα είδη, ενώ ε, την παλαμίδα την υποεκμεταλλευόμαστε. Να μην υπερεκμεταλλευόμαστε τα δύο, αλλά ίδια, ενώ την παλαμίδα την υποεκμεταλλευόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, γιατί είναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 22 ε, σκάφη από την Ισπανία, 16 από τη Γαλλία και 2 από την Ιταλία. και δύο ε, από την Ισπανία, δύο από τη Γαλλία και δύο από την Πορτογαλία, ε, την Παραγαδιάρικα. Είναι πολύ Σημαντικά επίσης ε, τα ψάρια τα οποία αποβιβάζονται στη Βικτόρια. Ε, επισκεφτήκαμε εκεί την πόλη, εντυπωσιαστήκαμε. μερικά μεταφορτώνονται, από τα ψάρια αυτά μεταφορτώνονται. Θέλουμε να εκφορτώνονται πολύ περισσότερα στην ε, Βικτόρια γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται εκεί και έχουν καλή απασχόληση. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση ε, πληρώνουμε 38.500 ε, ε, τα πρώτα χρόνια και 52.000 ε, για τις άδειε τα τελευταία χρόνια για τα σκάφη. Εγώ θέλω το, επίσης τα ψάρια να εκφορτώνονται όσον τον περισσότερο στις Σεϊχέλες. Δεν θα μιλήσω για την πειρατεία. Είναι πραγματικά τρομακτικές μερικές από τις ιστορίες που ακούσαμε για τους πειρατές. Αλλά γενικά όπως και, να κρίνουμε την κατάσταση, τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα παλιά, παρά παλιότερα. Φυσικά πρέπει να καταδικάσουμε την ε, πειρατεία με τους πιο ισχυρούς όρους. Ίσως θα πρέπει να αφιερώσουμε και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο σημείο στην έκθεση όπου ρητά να καταδικάζουμε την πειρατεία. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαγκερ για το θέμα της πειρατείας. Η Κομισιόν μπορεί να μας πει πότε έγινε η τελευταία επίθεση πειρατών με επιτυχία 18 μήνες πριν από τότε που άλλαξε το πρωτόκολλο ούτω ώστε ε, μπορούν να από ελικόπτερα τώρα οι στρατιωτικοί να πυροβολούν το μοτέρ του του αλλιευτικού σκάφους για να σταματήσει, του πειρατικού αλλιευτικού δηλαδή. Γιατί δεν έχει νόημα ας πούμε, να προσπαθούμε από την ακτή να πυροβολήσουμε αυτά τα σκάφη. Τώρα από ελικόπτερα είναι δυνατόν μετά την αλλαγή του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Πατράου Νέβε, την εισηγήτρια, για την ποιότητα της εκθεσή τη και για την πληρότητα των πληροφοριών τη. Να ξεκινήσω από κάποιες, απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις που μου τέθηκαν από του ευρωβουλευτές. Καταρχά για το θέμα των καρχαριών. Το συζητήσαμε τελευταία φορά. Ε, Εκπλήσω με τα νούμερα που αναφέρετε. Γιατί για μας είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με, με την αλήψη καρχαριών. Ε, η έκθεση αξιολόγησης λέει άλλα νούμερα. Ένας, βέβαια, μιλάει συνολικά για τον Ινδικό ε, ωκεανό. 4% των παρεμπιπτών των αλίευμάτων είναι καρχαρίες. Ε, και το 2% από αυτά δραπετεύουν ζωντανά. Δηλαδή, ουσιαστικά, είναι μικρός ο αριθμός των καρχαριών που, που ψαρεύονται κατά λάθο στον Ινδικό ωκεανό. Και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, μια και τα παραγαδιάρικα δεν είναι ενεργά και έχουμε ουσιαστικά γρηγροί που είναι, δραστηριοποιούνται εκεί, ο κίνδυνος ε, να ψαρέψουμε καρχαρίες κατά λάθο είναι ακόμα μικρότερος. Δεν υπάρχει ποσόστοση πάντως στα, στα πλαίσια των διατάξεων του πρωτοκόλλου αυτού. Τώρα, για τον εξοπλισμό συγκέντρωσης ηχθείων, Σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι εξοπλισμοί από ένα τμήμα του στόλου. Υπάρχουν μέτρα διαχείρισης, υπάρχει μια πλαισίωση αν θέλετε για αυτό τον εξοπλισμό στα πλαίσια της ε, σύμβασης ε, του Ινδικού ωκεανού για την ε, αλίευση των θηνοειδών. Οι ίδιοι επαγγελματίε θέλουν να δημιουργήσουν εξοπλισμούς πολύ πιο οικολογικούς και που αποφεύγουν τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα κάποιων ε, ηχθείων, κυρίως χελωνών. Τέλος πάντων, τους εξοπλισμούς αυτούς τους επιτρέπουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, το επιτρέπουν και οι Σεχέλες επίσης με, στην νομοθεσία τους να, να χρησιμοποιούν οι ψαράδες τέτοιου εξοπλισμούς. Για την τομεακή ενίσχυση, σημαντικό στοιχείο αυτού του πρωτοκόλλου. Πρέπει να υπενθυμίσουμε, όπως έκανε και η ότι μειώνουμε την ε, παρουσία μας και την πρόσβασή μας και πληρώνουμε λιγότερα εκεί για την ε, πρόσβασή μας στα νερά της, αλλά αυξάνουμε την ε, στήριξη του τομέα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία υποφελούνται άμεσα από την στήριξη της μικρής κλίμακας αλίας. Ούτως ή άλλως γενικά η αλία συνεισφέρει πάρα πολύ στο σύνολο της οικονομίας ε, των Σεχελών και επομένως στηρίζουμε τον τομέα. Είναι βασικό στοιχείο για να ενισχύσουμε την ε, διαχείριση της αλίας σε τοπικό επίπεδο και να ενισχύσουμε την αποδοχή της παρουσίας μας από τον πληθυσμό και τους ενδιαφερόμενους στις Σεχέλες. Επίσης, επευκαιρία να σας πω ότι μια μεικτή επιτροπή θα οργανωθεί το Μάρτιο, στις 24 Μαρτίου, αλλά θα επιβεβαιωθεί αυτή η ημερομηνία. Θα σα ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Θα είναι η πρώτη μεικτή επιτροπή για το πρωτόκολλο αυτό. Και ο στόχος της θα είναι να συμφωνήσει για το πρόγραμμα που, αφορούν, που αφορά την στήριξη του, του τομέα τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για ένα πολυετές πρόγραμμα με διάφορες δράσεις, διάφορους δείχτες που θα επιλεγούν ανά έτος. Αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν ε, με διάφορες υποδομές, κυρίως την ε, ε, οικοδόμηση ενός νέου, μιας νέας, ενός νέου κυματοθράφτη που θα χρησιμοποιηθεί και από τους αλείς. Ενίσχυση των μέτρων ελέγχου και εποπτείας επίσης και ενίσχυση του δυναμικού κυρίως κατάρτιση των ανθρώπων που δουλεύουν στην αλληλεία και των ε, ψαράδων που μπαίνουν στα ληφτικά σκάφη. Ε, σήμερα υπενθυμίσαμε τις οικονομικές επιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο την αλία αλλά και τις λιμενικές δραστηριότητες αλλά και το γεγονός ότι μπαρκάρουν ναυτικοί και έτσι μαθαίνουν οι ντόπιοι την αλία και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο του πρωτοκόλλου. Αυτά για την τομεακή στήριξη. Θα σας ενημερώνω βέβαια τακτικά για την χρησιμοποίηση που γίνεται από τις Αιχέλες αυτής της τομεακής στήριξης, λογικό είναι να το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την πειρατεία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το θέμα της πειρατείας. Είναι ένα ζήτημα που υπεύθυνοι είναι διάφοροι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και η Επιτροπή εξωτερικής δράσης. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε Ιχέλης βελτιώθηκε η κατάσταση πολύ. Υπάρχουν διάφορα μέτρα πρόληψης και αποτροπής που δημιουργήθηκαν ε, και που χρησιμοποιούν και τα δικά μας σκάφη με μηχανισμούς διαφορετικούς, με άλλα μέτρα χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, άλλα οι Ισπανοί. Μερικές φορές έχουμε στρατιωτικούς, μερικές φορές έχουμε ιδιωτικούς σεκιουριτάδες. Σχεδόν η πειρατεία όμως ε, εξαφανίστηκε από την ΑΟΖ της, ε, των Σεχελών. Δεν έχω την τελευταία ημερομηνία τώρα που συνέβη το τελευταίο κρούσμα πειρατείας, αλλά διαπιστώνουμε μια βελτίωση Εντυπωσιακοί συμφωνούν όλοι οι φορείς επιτόπου. Ε, επί χρόνια χρηματοδοτήσαμε ένα σχέδιο ελέγχου επισκόπησης του Ινδικού. Θα συνεχίσει η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, όχι από το Ταμείο ΜΑΡΕ. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα μέτρα, όλα τα μέσα μάλλον που έχουν οι πέντε χώρες τέρι ε, στην περιοχή για να καταπολεμήσουμε και την πειρατεία αλλά και την παράνομη λαθρέα και άναρχη Νομίζω ότι είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Κατά τα άλλα, να μην επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν τελευταία φορά. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ που διευκρινίσατε ότι είναι καλύτερη συμφωνία για σας από την προηγούμενη. Υπάρχει διαφάνεια, εφαρμόζει διάφορες αρχές της μεταρρύθμισης, ε, μια κατάρτιση για τους ε, που παρέχουν οι πλειοκτήτες. Επίσης, πληρώνουμε με βάση το τι ψαρεύουμε πραγματικά. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχουν διάφορες προσαρμογές οι οποίες έγιναν σε αυτό το νέο πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό αλίευσης, τον, ε, τις ποσότητες αναφοράς και λαμβάνουμε υπόψη μας την ε, χρήση που κάναμε στο πρωτόκολλο του στο παρελθόν. Η παρουσία μας Πρέπει να σας πω μάλλον ότι τα λεφτά που πληρώνουμε είναι λιγότερα. Από 5,6 εκατομμύρια πάμε ε, στα 5,3 για τα 5 χρόνια και μετά στα 5 για τα δύο τελευταία. Ε, η κυρία Πατράου Νέβες για την τελική της παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλια που έγιναν δεν αφορούσαν τόσο πολύ τη δική μου παρουσίαση. Αφορούσαν πιο πολύ τις ε, διατάξεις συγκέντρωση ηχθείων κλπ. Η Κομισιόν ήδη απάντησε. Υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Για το θέμα των καρχαριών ήδη το σχολίασα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ε, δεν γνωρίζουμε το επίπεδο βιωσιμότητάς τους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μόνο σε σχέση με την έκθεση ότι ζητούμε από την Κομισιόν να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα στοιχεία που έχει σε ό,τι αφορά τις μικτές τεχνικές συνεδριάσεις, τις, ε, ε, τα συμπεράσματα και τη, τα πρακτικά. Επίσης θέλουμε πληροφορίες για την, για την πρακτική στήριξη που παρήχαμε στον τομέα μέσω του πολιτικού προγράμματος σημαντικά στοιχεία για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας με αντικειμενικό και σοβαρό τρόπο. Στο σημείο 3 ζητούμε εκπρόσωποι της ε, Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις μεικτές ε, συνεδριάσεις, ε, τις αποκαλούμενες μικτές συνεδριάσεις. είναι σημαντικό να θεσμοθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την παρουσία. Και στο σημείο 4 ζητούμε στην τελευταία χρονιά ισχύω αυτής της συμφωνίας και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή της να διαθέτουμε ε, μια έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγηση τη λειτουργία συμφωνία, τόσο εμεί όσο και το Συμβούλιο, ε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ε, το πώ λειτουργήσε η συμφωνία αυτή για τον Ευρωπαϊκό Λευτικό Στόχο. Ε, στόλο, συγγνώμη. αυτά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία ζητούμε. Κυρία Λεβίνα έχει μια ακόμα ερώτηση νομίζω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Πατράο ε, έκανε την ίδια παρατήρηση την προηγούμενη φορά. Είπε δεν μπορούμε απλά να μιλάμε για καρχαρίες, θα πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα είδη καρχαριών. Και στην Επιτροπή Αλίας του Ινδικού Ωκεανού από ό,τι γνωρίζω απαγορεύεται η αλία τριών ειδών, η εκφόρτωσή τους, η πώλησή τους κλπ. Επίσης οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες και ο λευκός καρχαρίας είναι απαγορευμένα είδη. Ε, εκτός από ότι υπάρχει στο παράρτημα 1 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά είδη καρχαριών. Ε, τα νούμερα που ανέφερα προέρχονται από την έκθεση της κυρίας Πατράου, όπου μιλάει για 5% ξηφία και 24% άλλα είδη. Ιδιαίτερα καρχαρίες και ξηφίες. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιους καρχαρίες αναφέρεται εκεί, αλλά μιλάμε για την Αλληλεία, στην Ταϊλάνδη, Ομάν ε, και σε Ιχέλες. Αυτά βρίσκονται στην έκθεση της κυρίας Πατράου και ε, γι' αυτό έθεσα και την ερώτησή μου. Το 5% στην έκθεση οφείλεται στο ότι τα παραγαδιάρικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και ε, τα περιπτώτα αλλιεύματα είναι λιγότερο από 5% στα παραγαδιάρικα στον Ινδικό ωκεανό. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που έθεσα την ερώτησή μου. Εάν λοιπόν συνεχίζουμε να έχουμε έξι παραγαδιάρικα, και έχουν συγκρίσιμα παρεπίπτωτα αλλιεύματα με τα, τα υπόλοιπα σκάφη, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι και τα ποσοστά είναι παρόμοια με τα άλλα σκάφη και γι' αυτό έθεσα την ερώτησή μου. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο εδώ, αν έχει δίκιο η Επιτροπή ή αν έχει δίκιο η κυρία Πατράου σχετικά με το 5%. Δηλαδή είναι 5% παρεπίπτωτα λιεύματα ή 5% των συνελικών ελιευμάτων των παραγαδιάρικων στον Ειδικό ωκεανό. Θα ήθελα αυτό να διευκρινιστεί. Επίσης δεν κατάλαβα ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης για τις διατάξεις συγκέντρωσης ισχύων που αναφέρει η Επιτροπή μέτρα διαχείρισης μπορεί να αναφέρει κανείς χωρίς να αναφέρει τι είναι αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πατράου, σε ό,τι αφορά αυτή την έμονη ιδέα για τους καρχαρίες, θέλω να πω ότι ε, υπάρχει ένας συμβιβασμός όλων των ενδιαφερομένων ε, για, να, για τη μείωση των αλλιευμάτων. Ε, η, εξάρτητα από το τι ε, αλλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιείται ε, τα παραγαδιάρικα για παράδειγμα στις Αζόρες ε, έχουν μεγαλύτερα παραλιεύματα από τα γρήγορα από, τη, ε, τα είναι. Ε, οπότε και εδώ δεν έχουμε ε, παραγαδιάρικα όπως ξέρετε, είναι ελάχιστα. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι θέμα σημαντικό για να το συζητάμε. Υπάρχει συμφωνία για τη μείωση των παρελευμάτων και ήδη τα παρελιεύματα σε ό,τι αφορά τα γρηγρή είναι πολύ μικρότερα από ό,τι αυτά για τα παραγαδιάρκεια. Και έχουμε κυρίω ρίσει σε χέλε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, σημείο 7. Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις νήσους Κομόρες. Α, ε, ε τροπολογίες για το προηγούμενο θέμα ε, μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι στις 12, ε, για το σημείο 6, έτσι. 17 Φεβρουαρίου μέχρι το μεσημέρι οι τροπολογίες. Περνάμε σημείο από τα πρωτόκολλα Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομορών. Όπως θα θυμάστε, το Γενάρη, στη συνάντησή μας η Κομισιόν μας υπέβαλε την πρότασή της, μας παρουσίασε την πρότασή της, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σήμερα ο εισηγητής ο κ. Βαλέσα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο στόχος της συμφωνίας και του πρωτοκόλου είναι να διασφαλίσει τις αλλιευτικές ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό στόλο στο, για το πλεόνασμα που υπάρχει. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που επιφέρει προς τη αξία. Δεν νομίζω ότι είναι επίμαχο το θέμα. Μπορούμε να στηρίξουμε τη συμφωνία. Είναι προς όφελος ε, της, ε, προς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέχρι τώρα η εφαρμογή της συμφωνίας έχει στεφθεί με πτυχία. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες αλλιευτικής σύμπραξης που επιτρέπουν στον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλιεύει στα ύδατα των Κομορών από το 2005 και μετά. Το πρωτόκολλο που συζητάμε αυτή τη στιγμή εν μέρη έχει εφαρμοστεί, έχει εφαρμοστεί προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου. Προβλέπεται μία κοινή επιτροπή και θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας. Το κόστος της ανέρχεται σε 600.000 ευρώ το χρόνο και έτσι 42 παραγαδιάρικα μπορούν να αλλιεύουν στην περιοχή, συγγνώμη, 42 γρήγοροι και 22 ε, παρακαδιάρικα. Έκλεισε το μικρόφωνο το μίλητη. Μπορούν λοιπόν περισσότερα σκάφη να είναι παρόντα στην περιοχή, ωστόσο έχει μειωθεί ο αριθμός τους λόγω της πειρατείας που αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. Η κατάσταση της πειρατείας έχει βελτιωθεί τώρα, ωστόσο παραμένει πιο δύσκολη η κατάσταση τώρα από ό,τι ήταν πριν το 2005. Πιστεύω ότι το πρωτόκολλο θα ωφελήσει και τα δύο μέρη δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν αντιρρήσεις. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλέσα. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς εσάς και προς την Κομισιόν. Ε, στη Μαγιώτα επικρατεί πολύ δύσκολη ε, πολιτική κατάσταση σε σχέση με τις Κομόρες. Ε, ανήκει στην Γαλλία, είναι μία από τις ε, υπερπόντιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλληλείς της Μαγιότ μπορούν να ωφεληθούν από την συμφωνία αυτή. Μιλάμε για αλληλεία μικρής κλίμακας Έχετε μιλήσει με τους αλληλείς, ε, ρωτώ την Κομισιόν, υπάρχουν επαφές, διότι νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή. Θα ήθελα πολύ να γνωρίζω πώς χειριζόμαστε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λοβέν, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή, καθότι μιλάμε για την ίδια περιοχή. Θα δράξω την ευκαιρία να ξαναρωτήσω την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα διαχείριση των διατάξεων συγκέντρωση ηχθείων, των ΦΑΤ. Εδώ μιλάμε για 20 παρακαδιάρικα και όπω είπε και η κυρία Πατράο, τα παρακαδιάρικα έχουν τα περισσότερα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα διαφόρων ειδών καρχαριών και εξηφίων. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα για να αποφύγουμε τα παρεπίπτωτα λιεύματα και καθότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα πέντε είδη που σας ανέφερα πριν, τα οποία είναι απαγορευμένα είδη, τον σφυροκέφαλο, τον λευκό καρχαρία, ε, καθώς και το σκυλόψαρο. Ε, ε, θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται όσον αφορά αυτά τα είδη. Θα δώσω το λόγο και ε, στους υπόλοιπους βουλευτές. Κυρία Πατράου, ζήτησα το λόγο για να υπογραμμίσω ότι αυτή και η προηγούμενη συμφωνία, όσο και, της Μαδαγασκάρ, και η συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη και τη Μοζαμβίκη επίσης, είναι συμφωνίες ε, σημαντικές για να εγγυηθούμε την παρουσία μας στην, ε, στον νοτιοδυτικό Ινδικό. Και όταν δεν είμαστε εμείς εκεί, ε, είναι κάποιοι άλλοι. η απουσία μας, η απομάκρυνση μας από ορισμένε περιοχές, για παράδειγμα εξαιτία της πειρατείας, βλάπτει τον στόλο μας. Δεδομένης της ε, σημασίας αυτών των ε, συμφωνιών για την ε, οικονομική βιωσιμότητα όχι μόνο της αλληλευτικής δραστηριότητας Ε, αλλά και, μια, και για μια γενικότερη ε, οικονομική δυναμική που περιλαμβάνει και πολλές έμεσες θέσεις απασχόλησης. Αυτές λοιπόν οι εκθέσεις θα πρέπει να ειδωθούν στο σύνολό τους. και ε, να ενταχθούν στην προβληματική της γενικότερης παρουσίας μας σε μια αλληλευτική ζώνη. Οι κανόνες μάλιστα οι οποίοι τηρούνται και γίνονται σεβαστοί είναι αυστηρότεροι σε σχέση με οποιαδήποτε παρουσία σε άλλη αλληλευτική ζώνη. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην Κομισιόν στον κύριο Μπέρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Στον εισηγητή μάλλον για την έκθεση αυτή που προτείνει να επικυρώσει, να συμφωνήσει το, το Κοινοβούλιο ε, το πρωτόκολλο αυτό για τις Κομόρες. Για το καθεστώς του Μαγιότ. Όταν διαπραγματευόμαστε αλληλευτικές συμφωνίες μας δεν κάνουμε πολιτική. Προσπαθούμε να ξεχερσώσουμε το έδαφος και να ξεπεράσουμε τις περισσότερες δυσκολίε που υπάρχουν. Οι αλληλευτικές ζώνες ε, ορίζονται αποκλείοντας τη ζώνη της Μαγιότ που είναι γαλλική επικράτεια. Ε, παρότι οι κομόρες ε, διεκδικούν τη Μαγιότ. Εμείς πάντως το ορίσαμε έτσι, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αφησιμίε, ούτως ώστε να μην δυσκολέψουμε του αλείς μας. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να υποθεί. Εν συνεχεία, οι αλείς της Μαγιότ έχουν ε, κυρίως μια μικρή κλίμακα αλεία που ανήκει πλέον στην αλεία, στον αλληλευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν σκάφη, δηλαδή, τα οποία είναι καταχωρημένα στη Μαγιότ που μπορούν να ψαρεύουν στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας και επομένως μπορούν να πηγαίνουν, χάρη σε αυτή τη συμφωνία, να ψαρεύουν τώρα στις Υπάρχουν πέντε γρηγροί, τα οποία είναι καταχωρημένα με σημαία Μαγιότ και τα οποία θα ανήκουν πλέον στον Ευρωπαϊκό Στόλο και θα μπορούν να ψαρεύουν στι Κομόρες στα πλαίσια αυτή τη συμφωνία και στα πλαίσια άλλων συμφωνιών του Ινδικού Ωκεανού και έχουμε και έναν στόλο από παραγαδιάρικα πιο έτσι, ε, τα οποία μπορούν επίση να επωφεληθούν από τι αλληλευτικέ ευκαιρίε που προτείνει το πρωτόκολλο με τι Κομόρες, που προσφέρει το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο. Επανέρχομαι τώρα στο ερώτημα που τέθηκε για τους καρχαρίες. Όντω υπάρχουν διάφορα είδη καρχαριών. Κάποια είδη απαγορεύεται να τα ψαρεύουμε. Και αυτά, αυτή την απαγόρευση την εφαρμόσουμε και στο στόλο μας. Αποφασίζεται σε περιφερειακό επίπεδο και υπάρχει προφανώς και εντάσσεται και στο μηχανισμό του πρωτόκολλου. Θα πρέπει δηλαδή ο στόλος να έχει μέτρα επιλεξιμότητας ούτω ώστε να μην ψαρεύει αυτά τα απαγορευμένα είδη. Υπάρχουν και άλλα είδη όμως καρχαριών τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύουν. Επαναλαμβάνω όμως τα παραγαδιάρικά μας δεν είναι πολύ παρόντα εκεί, δηλαδή οι στόλοι δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. Άλλα κάνουν οι Ταϊβανοί, ας πούμε, και άλλα κάνει ο δικός μας στόλος. Δεν πρέπει ε, να κάνετε τέτοιες ε, συνδέσεις, διασυνδέσεις. Επίσης πρέπει να διακρίνουμε τα διάφορα είδη παραγαδιάρικων. Κάποια παραγαδιάρικα με ισπανική ή πορτογαλική σημαία, θεμητός πώς μπορούν σε κάποιες περιοχές να ψαρεύουν και καρχαρίες. Αν όμω λάβουμε υπόψη μα τα παραγαδιάρικα, τα γαλλικά του Ινδικού, με σημαία Μαγιότ ή Ρεϊνιό, ε, ψαρεύουν άλλα είδη. Έτσι. Ας πούμε, τα παραγαδιάρικα, τα γαλλικά, ε, ψαρεύουν κυρίως ε, ή τόνο. Ξυφία ή τόνο και όχι καρχαρία. Επίσης, ε, ο εξοπλισμός συγκέντρωση ηχθείων επιτρέπεται. Ε, και προβληματιζόμαστε αυτό το θέμα και σε επίπεδο περιφερειακό και ο κλάδος ε, ασχολείται και προσπαθεί να τα καταρτήσει πιο συμβατά με την διατήρηση των οικοσυστημάτων και των αποθεμάτων. Γίνεται συνέχεια βελτίωση αυτών του εξοπλισμών. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσετε αυτό το θέμα στα πλαίσια μιας έκθεσης που αφορά την αλία θηνοειδών και τη χρήση των ε, εξοπλισμών αυτών συγκέντρωση ηχθείων στην αλίευση θηνοειδών. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, θα μιλήσει ο κ. Βαλέσσα για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να σας καλέσω να υποστηρίξετε το πρωτόκολλο. Αν εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά, βλέπουμε σαφώς ότι τα υπέρ ξεπερνούν κατά πολύ σε αριθμό τα κατά. Και το βασικό ερώτημα είναι εάν η παρουσία του ευρωπαϊκού στόλου θα είναι καλύτερη από την απουσία του. Και κυρία Πατράου, νομίζω θα συμφωνήσετε με αυτήν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το πρωτόκολλο και τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 17 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, όπω και με την προηγούμενη έκθεση. Περάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 8. Παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β του ενημερωτικού σημειώματο με θέμα εσωτερική αλία και ΚΑΠ. Γνωρίζετε ότι ε, ζητήσαμε αυτή την, ε, αυτό το ενημερωτικό σημείωμα. Το ανέλαβε το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής το έχετε το ενημερωτικό σημείωμα, δεν πρόκειται να σας μιλήσω εγώ για αυτό, γιατί βρίσκεται παρούσα η κυρία Στεφανή Νιούμαν που το συνέταξε, είναι από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει το ενημερωτικό αυτό σημείωμα. 20 ε, λεπτά το πολύ παρακαλώ. Good morning. Um, Καλημέρα. Λέγομαι Στέφανη Νιούμαν. Δουλεύω για το Ινστιτούτο ε, Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και η Κομισιόν ε, μου είπε να σας κάνω μια ενημέρωση για την ε, πολιτική εσωτερικών υδάτων και την κοινή αλληλευτική πολιτική. Θα σας πω τα βασικά στοιχεία και στη συνεχεία θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Η ενημέρωση αυτή γίνεται για να μιλήσω για την εμπορική αλία, δηλαδή αποκλείουμε την, την ψυχαγωγική αλία και την αλία που γίνεται για, να, για επιβίωση. Επίσης, ε, ε, ελέγχουμε τον τομέα, τα είδη, την κατανομή, τις ληφτικές μεθόδους, τα αλλιεύματα, ε, την απασχόληση, μια επισκόπηση των αγορών και την κοινωνικο-οικονομική σημασία του κλάδου. Επίσης, αναλύει την επίπτωση της μεταρρύθμισης κοινής αλληλευτικής πολιτικής στην αλληλεία εσωτερικών υδάτων. Αναθεωρήσαμε την τεκμηρίωση. Ε, είδαμε εκθέσεις σε βάση δεδομένων και πολύ νωρίς καταλάβαμε ότι οι πληροφορίες για αυτή την αλία είναι πολύ ετερογενείς. Ε, δεν ε, συγκεντρώνονται στοιχεία τακτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η εμπορική αλία εσωτερικών υδάτων είναι διαφορετική από κρατός μέλος σε κρατός μέλος. Ε, Όμω δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τα δικά μα στοιχεία. Βασιστήκαμε στην πρόσφατη τεκμηρίωση που υπάρχει, στα στοιχεία που έχουμε για την αλληλεία αυτή. Τι είναι αυτή η αλληλεία, καταρχά. Είναι η αλληλεία που υπάρχει σε μεγάλες φυσικές λίμνες, σε ταμιευτήρες, δεξαμενές, α, α, λιμνοθάλασσες, εκβολές, ποταμό και ποταμούς. Ε, μιλάμε για μεταναστευτικά είδη του γλυκού νερού, ε, που περνάνε ένα τμήμα τη ζωή στο γλυκό νερό και ένα τμήμα στο αλμυρό νερό. Αυτά είναι τα διάδρομα ήδη θα τα λέμε. Ε, είναι κυρίως αυτά που ψαρεύουν οι, οι αυτοί. Ε, τα ψαρεύουν σε παράκτιες περιοχές, σε ποταμούς και κυρίως σε αυτές τις περιοχές τέτοια είδη ε, εκμεταλλευόμαστε. Βλέπουμε κάποια παραδείγματα στα slides. Από πάνω, αριστερά, έχουμε την πέστροφα, ε, το ευρωπαϊκό χέλι, τον ξύριγχο, Αυτά είναι τα βασικά είδη. Είναι διάδρομα είδη και εστιάζουμε, θα επίσης πολύ στα διάδρομα είδη και στο χέλι. Για τον όγκο τώρα των αποθεμάτων. Κυρίως ε, τα ψάχνουμε στα γλυκά νερά. Ε, είναι κυπρινοειδή, Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Το ΚΑΡΠ, ε, το ποταμολάβρακο, το χέλι. Πού, πού, υπάρχουν, ε, πού υπάρχει αυτή η αλληλεία. Υπάρχει σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη. Βέλγιο, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία. Αυτά τα κράτη δεν έχουν τέτοια εμπορική αλληλεία εσωτερικών υδάτων. Στη Δανία, στην Τσεχία, και στην Κροατία, ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Λιγότερο από 30 άτομα ασχολούνται. Στα υπόλοιπα 19 κρατη αυτή η αλία είναι σημαντική με τουλάχιστον 100 αλίες που ασχολούνται εκεί. Θα σας μιλήσω για τα διάδρομα ήδη και το ευρωπαϊκό χέλι. Ε, το μικρό χέλι επίσης που είναι κυρίως στην ακτή του Ατλαντικού, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και στο κανάλι της Μάχης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πώς κρατάμε σε καλά επίπεδα αυτά τα ψάρια ε, με την ανασύσταση των ειδών που εισάγονται εισάγουμε νέα είδη από άλλες χώρες. Λοιπόν, ε, μέθοδοι και εργαλεία. Υπάρχουν 14 με 15.000 ε, αλληλευτικά σκάφη στα, στον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εκτίμηση είναι πολύ χοντρική, με βάση τα όσα λένε οι πυρογνώμονε. Όλα τα κράτη-μέλη δεν απαιτούν να καταχωρούνται αυτά τα σκάφη. Μερικά, τα περισσότερα από αυτά είναι μικρότερα από 8 μέτρα και έχουν 30 ε, ύπου στο μοτέρ. Δεν χρησιμοποιούν επίσης ενεργά ε, αλλιευτικά εργαλεία, αλλά δρανή. 14.000 σκάφη λοιπόν, να δούμε. Είναι το 14% του συνολικού ευρωπαϊκού ε, στόλου. Και μοιάζει βεβαίω η αλία αυτή ε, με την ψυχαγωγική αλία και την αλία μικρής κλίμακας στα θαλάσσια ύδατα. Συνολικά, τα δρανή εργαλεία χρησιμοποιούνται κυρίως για αυτή την αλία. Παγίδες, ε, πετονιές, ε, δίχτυα, αδρανή, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Ε, σε μεγαλύτερα ύδατα, σε μεγάλες ας πούμε λίμνες και σε, σε δέλτα χρησιμοποιούνται ενεργά εργαλεία. Στην Εστονία που ψάχνουμε ποταμολάβρακο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη Βόρεια Ιρλανδία Επίσης στις λίμνες της Άλπης που ψαρεύουμε ε, χέλη, επίσης χρησιμοποιούμε πιο έντονα εργαλεία. Πέρα από τα 14.000 σκάφη υπάρχουν επίσης περίπου χίλιοι ψαράδες που ψαρεύουν από την ακτή ή ψαρεύουν από, πάνω, από τον πάνω τον πάγο, ας πούμε, στην Εστονία, στην Φιλανδία. Το χειμώνα. Για τα αλλιεύματα. Ετήσια είναι περίπου 35.000 τόνοι με βάση εθνικές στατιστικές και τα όσα λένε οι Δηλαδή, ποιο είναι το πλαίσιο. Είναι περίπου το 1% των συνολικών αλλιευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2008 αυτά. Είναι σαφές ότι η συνεισφορά της αλίας στην συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή είναι αμεληταία αλλά είναι μέσος όρος και η συνεισφορά εθνικές, στην εθνική παραγωγή μερικές φορές ε, για λίγα κρατημέλη είναι πολύ σημαντική. Στη Ρουμανία, ας πούμε, ε, έχουμε 89% ψάρια γλυκού νερού. Στη Βουλγαρία είναι 13%. Φυσικά σε περίκλειστα κρατημέλη η αλληλεία εσωτερικών υδάτων είναι το 100% της συνολικής παραγωγής ηχθείων στη χώρα. Η Φιλανδία έχει τα ψηλότερα αποθέματα, ψάρεματα. Ρουμανία η συνεχεία. Ιταλία. 4.398 τόνοι, 4.284 τόνοι για τη Ρουμανία και 3.915 για την Ιταλία. Γύρω στα 100 με 110 ε, εκατομμύρια ευρώ έχουμε στην Ευρώπη αυτό είναι το 1 με 2% της αξίας όλων των εκφορτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μικρό ποσοστό. Πέντε κράτη-μέλη ε, είναι το, ε, δίνουν Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Φιλανδία και Ιταλία ε, αποτελούν το 50% των συνολικών εκφορτώσεων αυτής της αλληλείας. Τώρα η απασχόληση στον κλάδο. 17.100 ψαράδες ψάρευαν το 2008-2009. Οι περισσότεροι όμως δούλευαν part-time. Ε, λόγω του ότι έχει εποχιακό χαρακτήρα αυτό το επάγγελμα, συνολικά αυτοί οι ψαράδες ε, στα ποτάμια και, στους, στα δέλτα των ποταμών ε, είναι περισσότεροι. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα διάδρομα ήδη ψαρεύονται εκεί. Και τα ψάρια που ψαρεύουμε στις λίμνες λοιπά είναι περίπου το 5%. Αλλά στις, ε, μόνο το 1 τρίτο των ψαράδων ψαρεύει σε λίμνες, μακριά από ποτάμια και δέλτα. Τώρα, για τα νούμερα απασχόλησης. Τα, οι 17.000 αυτές ψαράδων είναι περίπου το 10% των συνολικών ψαράδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές ξεχνάμε τη σημασία του κλάδου σε κάποια κράτη-μέλη βέβαια με αυτά τα νούμερα. Στη Ρουμανία είναι περίπου το 90% και στη Φιλανδία το 60% ε, των ψαράδων, αυτοί που ψαρεύουν δηλαδή ε, στα εσωτερικά ύδατα. Τώρα οι αγορές για τα ψάρια γλυκού νερού. Τα περισσότερα ψάρια πηγαίνουν στην περιφερειακή εθνική αγορά μέσω χονδρέμπορων ή με, μέσω άμεσης ε, πώληση στους ιδιώτες, με εξαίρεση την Εστονία, όπου το ποταμό ε, δίνεται στους μεταπίτες και μετά εξάγεται στον ε, Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μικρό χέλι ε, το εκμεταλλευόμαστε και πουλιέται και σε άλλα και διεθνώς. ότι περιορίστηκε αυτό το διεθνές εμπόριο μετά από μια απαγόρευση το 2009. Για να συνοψίσω όλα όσα είπαμε στιγμής, να δούμε τις επιπτώσεις των αριθμητικών στοιχείων. Υπάρχει δυσανάλογος αριθμός ε, ψαράδων που απασχολείται εκεί σε σχέση με την παραγωγικότητα, μόνο το 1% της ευρωπαϊκής παραγωγής δηλαδή. Και αυτό οφείλεται στο ότι πολύ, έχει πολύ ένταση εργασίας αυτή η μορφή αλίας αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες αξίες στον κλάδο, η ψηλή απασχόληση, την ανέφερα ήδη. Τα περισσότερα ψάρια όμως που ψαρεύονται εκεί, στην πραγματικότητα καλύπτουν ε, συγκεκριμένες αγορές, την τοπική αγορά, την περιφερειακή αγορά. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν μεγάλη προσθέμενη αξία. Και επίσης ε, έχουν μεγάλη σημασία πολιτιστική και κληρονομική και με βάση την παράδοση. Η γνώση επίσης ε, παραδίδεται από γενιά σε γενιά, επομένως η σημασία της αλίας αυτής πολιτιστικά είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδεχομένω και περιβαλλοντικά. Οι επαγγελματικές οργανώσεις στον κλάδο τώρα. Από ό,τι φαίνεται, η εμπορική αυτή αλία έχει πρόβλημα εκπροσώπησης. Μόνο στη Φιλανδία και στη Γαλλία έχουμε επαγγελματικές οργανώσεις, ειδικά για αυτούς τους ψαράδες. Σε άλλες χώρες η εμπορική αλία εσωτερικών υδάτων ε, εκπροσωπείται από οργανώσεις που συμπεριλαμβάνουν και τις υπόλοιπες μορφές αλίας, την αναψυχή, την ψυχαγωγική, Τη μικρή κλίμακα κτλ. Είναι μειονότητα λοιπόν και επομένω τα συμφέροντά του συχνά παραβλέπονται. Ορισμένοι λένε ότι ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των αλλιέων και έλλειψη πόρων είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει τέτοια εκπροσώπηση. Και γι' αυτό οι αλλοί αυτοί και οι αλλοί ε, δεν μπορούν να εφαρμόσουν ούτε για λόγους α, πώλησης, ούτε για την αγορά ούτε για την εκπροσώπηση, ε, συνολικές στρατηγικές. Σας παρουσίασα συνολικά τον κλάδο, όσο έχει σήμερα. Και τώρα θα εξηγήσω λιγάκι που εντάσσεται στην πολιτική, την αλληλευτική, ο κλάδος αυτός. Η αλληλεία αυτή τη χάνει διαχείριση ε, στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας. Εμείς δεν έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες για αυτή την αλληλεία. Ε, παρότι υπάρχουν και τα διάδρομα ίδια αυτά, τα οποία περνάνε από το ένα νερό στο άλλο. Ε, και η διάκριση ε, οικολογικός πώς δεν είναι σωστή. Ούτε για τη διατήρηση των ειδών, ε, δεν αντιμετωπίσουμε συνολικά τον κύκλο ζωής των ειδών, αλλά έτσι έχει εξελιχθεί η συν το χρόνο. Είναι σημαντικό να σας αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία που επηρεάζουν τη διατήρηση των ε, ε, ειδών των φρέσκων, των γλυκών νερών και των διατημάτων τους η οδηγία πλαίσιο για το νερό, η οδηγία για τα ενδιατήματα και η οδηγία, ο κανονισμός, συγγνώμη, life. Για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Συνολικά, η αλλή αυτή δεν υπόκειται στους κανόνες κοινή αλληλευτικής πολιτικής, όμως ισχύουν για, την, για τα διάτρομα είδη στο θαλάσσιο τμήμα της ζωής τους. Ένα παράδειγμα είναι στο Βόρειο Ατλαντικό. Τα κυρίαρχα κράτη έχουν το ρόλο τους ε, για τη ρύθμιση της ε, αλίας του ε, Σολομού στα ποτάμια τους και δεν μπορούν να ψαρεύουν σε περιοχές που δεν είναι της επικράτειάς τους και πέρα από τα 12 μίλια τους. Αντίθετα, στη Βαλτική η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την αλία του Σολομού μέσω ΤΑΚ και ποσοστώσεων. Και τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, εθνικά μέτρα μόνο στα ποτάμια τους. Το ευρωπαϊκό χέλι υπόκειται σε μακροπρόθεσμο σχέδιο διατήρησης. Υπάρχει λοιπόν μια πλειάδα προσεγγίσεων για τα διάφορα είδη. Για το Σολομό της Βαλτικής τώρα, τον διαχειριζόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τάκ ποσοστώσεων, κλειστών ε, εποχών, ε, περιορισμών στα ληφτικά εργαλεία και έχουμε εθνικά μέτρα στα ποτάμια. Το 2011 ένα πολιετές πρόγραμμα διαχείρισης προτάθηκε από την Κομισιόν για αυτό το Σολομό που θα καλύπτει και τη θάλασσα και τους ποταμούς. Ε, καλύπτει όλο τον κύκλο μετανάστευσης του Σολομού. Ε, υπάρχει μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και οικονομική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την ανασύσταση του πληθυσμού μέχρι το 2015. Έχουμε υψηλού στόχους αναπαραγωγής, αυστηρότερους ε, κανόνες για την ανασύσταση του αποθέματος στα ποτάμια. Αυτό πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν συμφώνησαν τα τρία, τα τρία θεσμικά όργανα για αυτά τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Το ευρωπαϊκό χέλι είναι πιο τυχερό, έχει ένα σχέδιο διαχείρισης και ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα πλαίσιο για την προστασία και την ε, βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού. Επίσης, σε ποτάμια, ε, σε ποταμόκολπους, ε, δέλτα κτλ. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν δεξαμενές ποτάμιες για να καλύψουν, για να προστατεύσουν το χέλι, να μειώσουν ε, την ανθρωπογενή ε, θνησιμότητα και να αυξήσουν τη διαφυγή του χελιού στη θάλασσα. Μία επισκόπηση της ε, εφαρμογής του σχεδίου από την ISIS πέρυσι δείχνει ότι τα δύο τρίτα των μέτρων που προτείνουν τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμοστεί. Τα μισά από αυτά ήταν μέτρα παρακολούθησης. Και τα μισά ήταν μέτρα περιορισμού της εμπορικής και, αναψυχα... και ψυχαγωγικής αλίας. Και το 1 τρίτο είχε εφαρμοστεί μερικώς ή καθόλου. Είναι συχνά μέτρα που αφορούν την ανασύσταση των ε, ενδιατημάτων, την, ανασ... την ανασύσταση του αποθέματος κτλ. Πάμε τώρα στη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και το βασικό κανονισμό αυτή η αλία δεν ρυθμίζεται από το βασικό κανονισμό της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Επομένως, γενικά δεν εξάρτηται από αυτόν. Με εξαίρεση τα διάδρομα ήδη, όπου εκεί η κοινή αλληλευτική πολιτική παίζει κάποιο ρόλο, ε, το ευρωπαϊκό χέλι και το σολομό της Βαλτικής, ε, η μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής είναι να φτάσουμε τα ίδια αυτά σε επίπεδο πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, να εφαρμόσουμε τα πολιετή προγράμματα και υποχρεώσεις για την εκφόρτωση και τα αποθέματα και τις, συγγνώμη, και τις απορρίψεις. Αν μεταρρυθμίσεις αυτές ε, εφαρμοστούν έγκαιρα και σωστά, δηλαδή για το Σολομό της Βαλτικής, αν εφαρμοστεί γρήγορα, και να έχουμε ποσοστά εκμετάλλευσης με βάση τις επιστημονικές συμβουλές μπορεί να υπάρξει ένα καμψί των ε, αποθεμάτων και να είναι βιώσιμος ο τομέας. Δυστυχώς οι επιδόσεις για την εφαρμογή ήταν ε, μάλλον κακές. Η οθέτηση των μακροπρόθεσμων σχεδίων διαχείρισης υπό την προηγούμενη πολιτική ήταν ε, αργή. Είχαν τσακωμούς τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους, διαφωνίες η μεταρρύθμιση του 2012 δεν καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα μέσω το οποίο τα πολιετή προγράμματα πρέπει να υιοθετηθούν. Υπάρχει κίνδυνος ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι τροχοπέδι στην εφαρμογή. Επιπλέον, όπου είναι δυνατόν, η ISIS χρησιμοποίησε το στόχο του MSY, δηλαδή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, που βασίζεται σε επιστημονικέ συμβουλέ, βέβαια. Το Συμβούλιο συχνά καθορίζει τάκ σε επίπεδα που ξεπερνούν αυτές τις προτάσεις. Στη πρόσφατη συνάντηση του Συμβουλίου έκαναν το ίδιο. Έβαλαν ε, τάκ για το σολομό της Βαλτικής πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των απορρίψεων, ε, για το σολομό της Βαλτικής έχουμε επίπεδα απορρίψεων 5 με 8%. Δεν είναι τεράστιο το ποσοστό, αλλά αρκετά σημαντικό παρόλα αυτά το σχέδιο απόρριψή των ε, απορρίψεων μπορεί να βοηθήσει την βελτίωση του αποθέματο του Σολομού, αλλά αν συνδυαστεί με άλλα μέτρα για να μειώσουμε την θνησιμότητα και τα επίπεδα τα ποσοστά συγγνώμη θνησιμότητας. Ο βασικό κανονικό έχει περιορισμένη αρμοδιότητα για την ε, αλία εσωτερικών υδάτων. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μέτρο ε, στα πλαίσια του Ταμείου για να υποφεληθεί η εμπορική και ψυχαγωγική αλία εσωτερικών υδάτων, με βάση μια πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν για αυτή την αλία δεν είναι πολύ σημαντική. Το προτινόμενο άρθρο για να υποστηρίξει αυτή την αλία είναι το άρθρο 42 το οποίο μοιάζει με το άρθρο που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Λιευτικό Ταμείο, EFF. Με τη διαφορά ότι έχουμε ε, δεν έχουμε υποστήριξη για την προσωρινή πάυση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και υπάρχει υποστήριξη ε, για τα σκάφη, ε, τον εξοπλισμό τους κτλ. Και, και την α, το να χρησιμοποιηθούν ε, τα σκάφη για άλλες δραστηριότητες. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πολλά, τα, πολλά κρατημέλη αυτό το μέτρο, μόνο εννέα. In Περισσότερη υποστήριξη προτείνει η Κομισιόν για την ανάπτυξη στρατηγικών, δικτύωση μεταξύ των τοπικών ομάδων, ε, ενισχύει την σημασία της δικτύωσης, προσπαθεί να πείσει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τα, τους του τους με ομάδες στήριξης, να αυξήσει την άμυλα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών ομάδων δράσης των αλλιέων και προσπαθεί να εισάγει την ευκαιρία πολλαπλής χρηματοδότησης, ούτως ώστε οι τοπικές ομάδες να έχουν χρηματοδότηση από πολλά, ε, πολλές πηγές. Με μία μεθοδολογία, κοινή μεθοδολογία για όλες τις αιτήσει, για όλα τα ταμεία, ούτως ώστε να είναι η χρηματοδότηση και συνεπής και συντονισμένη. Επίσης ε, υπάρχουν ε, σημαντικά κίνητρα. Ε, το ποσοστό χρηματοδότησης αυξήθηκε σε 75%. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της μεταρρύθμισης? Τα προτινόμενα μέτρα για αυτή την αλληλεία δεν άλλαξαν πολύ. Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι τόσο σημαντική για την αλληλεία εσωτερικών υδάτων, όσο για τη θαλάσσια αλληλεία, γιατί ουσιαστικά η μέθοδοι αλλίευσης είναι αδρανή αλλιευτικά εργαλεία γενικά και ουσιαστικά είναι οι πιο βιώσιμες ε, μέθοδοι, ε, χρησιμοποιούν μικρή, μικρά ποσοστά ενέργειας ούτως ή άλλως, καταναλώνουν λίγη ενέργεια, επομένως το EMFF έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτή την αλληλεία για να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση των κοινοτήτων που στηρίζονται από αυτή την αλληλεία. So, to conclude, um, Κλείνοντας, αυτή η αλληλεία εκφεύγει τη αρμοδιότητα κοινή αλληλευτική πολιτική και δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη μεταρρύθμιση του βασικού κανονισμού με την εξαίρεση των διάδρομων ειδών. Η κοινή αλληλευτική πολιτική μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατάσταση του Σολομού της Βαλτικής και του Ευρωπαϊκού Χελιού ενδεχομένως. Αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Μέσω ε, Μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας, ε, που υποστηρίζει ε, δραστηριότητες σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτής της αλίας. Πολύ ωραία. Έχει το λόγο και ο Στίβενσον καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Είπατε στην αρχή της παρουσίασής σας ότι θα αναφερθείτε και στην ηχθειοκαλλιέργεια, μου φαίνεται πως άκουσα. Όχι. Ε, μάλλον το αντίθετο είπα, ότι ε, δεν θα αποτελέσει μέρος της παρουσίασής μου. Διότι αναρωτιόμουν αν έχετε κάνει κάποια μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της ηχθειοκαλλιέργειας του Σολομού στα άγρια αποθέματα Σολομού. Μήπως έχετε κάνει κάποια σχετική έρευνα. Επειδή το πεδίο εφαρμογή της ενημέρωσης ήταν περιορισμένο, ε, επικεντρώθηκα πιο πολύ στις άμεσες συνέπειες, αλλά καθότι η μεταρρύθμιση έχει ενθαρρύνει την ηχθειοκαλλιέργεια, υπάρχει ο κίνδυνος σε πολλά επίπεδα αυτό να αποτελέσει απειλή για την αλληλεία λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων όπως είναι η γενετική μόλυνση από τους καλλιεργομένους ηχθείες καθώς και ο ανταγωνισμός στην αγορά θα αποτελέσει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον, ωραία. Σας ευχαριστώ για αυτήν την απάντηση. Όσον αφορά το θέμα, το διοργανικό στο οποίο αναφερθήκατε. Το αδιέξοδο. Μπορεί να γνωρίζετε ότι δημιουργήθηκε μία task force στην οποία συμμετέχουν ε, τα θεσμικά οργάνα και έχουμε ήδη καταλήξει σε μία συμφωνία όσον αφορά τα ε, μεμονωμένα αποθέματα πελαγικών ειδών. Και η Κομισιόν είπε ότι θα ετοιμάσει πολυετή σχέδια για μεμονωμένα είδη πελαγικά. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να ισχύει και για τον Σολομό της Βαλτικής. Μπορεί λοιπόν να εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που το ακούω. Η κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή, η οποία επιβεβαίωσε την εικόνα που ήδη είχα σχετικά με την αλία εσωτερικών υδάτων που από ό,τι ε, γνώριζα ήταν μικρής κλίμακας θα ήθελα να θίξω ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Σουηδία. Για παράδειγμα, ότι στην λίμνη Γέλμαρεν, όπου οι αλλοίς πριν 10 χρόνια συγκεντρώθηκαν, ε, υπήρξε πρόβλημα υπεραλίευσης, αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν κάτι γι' αυτό, αύξησαν το ελάχιστο μέγεθος ε, ματιού, δεν θυμάμαι ακριβώς τα χιλιοστά, Επίσης το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης ε, των ψαριών που αυξήθηκε από τα 30 στα 50 εκατοστά. Έτσι κατάφεραν να αντιστρέψουν την όλη κατάσταση και κατάφεραν ε, να ε, να πιστοποιηθεί η αλή αυτή και σχεδόν βγάζουν εκατομμύρια κορώνες Σουηδίας. Τα καταφέρνουν πολύ καλά είναι λοιπόν ένα από τα λίγα παραδείγματα που βλέπουμε πώς μπορεί να αντιστραφεί ένας φαύλος κύκλος και να μην ανταγωνίζονται για το πώς θα πιάσουν τα μικρότερα ψάρια προτού τα πιάσει οποιοδήποτε άλλος, ε, του να συμφωνήσουν δηλαδή ε, να αυξήσουν το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Αλλά παρουσιάστηκε και ένα άλλο πρόβλημα, διότι για να διατηρήσουν την ε, πιστοποίηση του Marine Stewardship ε, Council πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των αλλιευμάτων. και οι Σουηδικές αρχές το κάνουν αυτό, αλλά μόνο στη θάλασσα και όχι κάθε χρόνο στις λίμνες. Και, και έτσι δεν ε, υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η πιστοποίηση. Το θέμα αυτό λύθηκε στη Σουηδία, τελικά έγινε η αξιολόγηση των αλλιευμάτων ε, και το θέμα. Τα λέω όμως όλα αυτά γιατί, διότι αποτελεί αυτό ένα παράδειγμα διότι λέγεται ότι δεν έχουμε καλή αξιολόγηση των αλλιευμάτων ε, στα εσωτερικά ύδατα. Στις λίμνες λοιπόν τα αποθέματα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τη στη θάλασσα, διότι αν το γνωρίζαμε αυτό θα ήταν χρήσιμο, διότι κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι πάντα θα πρέπει να κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπεραλίευση, αλλά εάν εξετάσουμε την κατάσταση των αλλιευμάτων στα εσωτερικά ύδατα, όπου η κάθε χώρα έχει τον έλεγχο. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε εάν όταν τα κράτη-μέλη έχουν την πλήρη αρμοδιότητα, αν μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα αλλιεύματα. Μια ερώτηση λοιπόν προς εσάς, εάν έχετε κάποια ιδέα σχετικά με ε, την κατάσταση των αλλιευμάτων στα εσωτερικά ύδατα και είναι σε καλύτερη κατάσταση ή σε χειρότερη τα αλλιεύματα αυτά από τη στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, βουλευτές και μετά ε, θα ακούσουμε τις απαντήσεις όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Νιούμαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, ιδιαίτερα η σχέση ανάμεσα στην αλία στη θάλασσα και την αλία εσωτερικών υδάτων η αλία εσωτερικών υδάτων σε πολλές χώρες ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και μάλιστα έχει και σημασία για τον τουρισμό στις χώρες αυτές. Όσον αφορά τα είδη όπως είναι ο Σολωμός και το Χέλη, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έχουμε ασχοληθεί εντατικά με τον κανονισμό του 2009 και το σχέδιο διαχείρισης ε, του χελιού εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, έχουμε καταλήξει και σε μια λογική λύση. Το ερώτημα είναι, επειδή μιλάτε για εξαγωγές μικρών χελιών και προϊόντων χελιού, η απαγόρευση εξαγωγής προς την Νοτιοανατολική Ασία, εκτός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνεχίζεται. Από πού ε, έχετε τα νούμερά σας, ε, πού γίνονται οι παραβάσεις, διότι είπατε κι εσείς ότι γίνονται εξαγωγές. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη με ερώτηση. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, έχετε στατιστικά σχετικά με τα, ε, με τα αρπακτικά πουλιά στις ε, λίμνες. Και... Έχουμε συζητήσει και το θέμα κάποιων ε, θηλαστικών που που τρώνε τα ψάρια, τι γίνεται και με την εραστεχνική αλληλεία το σχετικό άρθρο στο, στο, νομοθέτημα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε την αλληλεία μικρής κλίμακας και η Κομισιόν είναι παρούσα. Ελπίζω αυτό να αναφερθεί σαφώς και στις διατάξεις εφαρμογής. Είδα όμως τα πρώτα έντυπα για τις αιτήσει υποστήριξης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Πάνω από 100 ερωτήσεις πρέπει να απαντήσει ένας μικρός αυτοαπασχολούμενος αλίας. Ε, εξετάσεις υγείας της γιαγιάς του πρέπει να δείξει για να πάρει 200 ευρώ. Πρέπει να ασχοληθούμε εδώ στην Επιτροπή μας ε, το θέμα αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι απαραίτητο δεν ε, πρέπει να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Κυρία Νιούμαν, ε, μπορεί αυτό να ξεφεύγει από τον τομέα σας, ε, αλλά έχει να κάνει με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Η Κομισιόν είναι παρούσα, και θα της δώσω το λόγο πριν τον κύριο Πένα, τον κύριο Τρίτε, ξέρω, και μετά στην κυρία Νιούμαν βέβαια για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσουμε στο τελευταίο τελευταία ερώτηση μόνο. Έχετε απόλυτη ελευθερία, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν απαντήσουμε σε αυτή την τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμε σε ό,τι αφορά την έκθεση. Όπως είπε και η επιστήμον, κυρία Νιούμαν, η, η τελική εκδοχή ε, είναι επί επιτρέπει περισσότερες δραστηριότητες ε, από τη αρχική πρόταση της Κομισιόν. Ε, το καινούργιο ταμείο δηλαδή επιτρέπει ε, να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες στην καινοτομία ή στην εμπορία. Τώρα, για το πώς χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των μέτρων που επιτρέπονται αυτή τη στιγμή και πάλι για τα εσωτερικά ύδατα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και τα στοιχεία αυτά φτάνουν μέχρι το Μάιο του 2013 χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί 630 δραστηριότητες ε, σε παράκτη με προϋπολογισμό 6,7 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Το κοινοτικό κομμάτι δηλαδή της χρηματοδότησης. Ε, σχεδόν όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν σχέση με υποδομές κατασκευή νέων υποδομών ή βελτίωση αλλιευτικών υποδομών. Τώρα υπάρχουν και κάποια ελάχιστα μέτρα σε, που αφορούν εξυγχρονισμό αλλιευτικών σκαφών για ελιές εσωτερικών υδάτων, αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσά αυτά. Τώρα, αυτά τα 6,7 εκατομμυρία αντιπροσωπεύουν το 0,6% περίπου των συνολικών δραστηριοτήτων του Ταμείου και περίπου 0,25% του συνολικού ε, προϋπολογισμού για τις πιστώσεις οι οποίες έχουν ήδη καταναλωθεί. Αν συγκρίνεται αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία της έκθεσης που περιλαμβάνουν το, τη συνολική αξία ε, της ε, παράκτειας αλίας νομίζω ότι η χρησιμοποίηση του ταμείου είναι λίγο χαμηλότερη. Η χρήση του ταμείου από τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτά τα μέτρα είναι λίγο χαμηλότερο από το ποσό το οποίο αναφέρει η έκθεση. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο ε, και ούτε και αν τα κράτη-μέλη έχουν ε, πράττουν σωστά ή όχι. Η μια μέση χρηματοδότηση είναι 10.000 ευρώ. Φαίνεται μικρό το ποσό αυτό, αλλά αντιστοιχεί πάνω κάτω στο πόσο κοστίζει να αλλάξει κανείς ε, τον κινητήρα του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ποιοτικά είναι σημαντικό. και είναι δύο με τρεις φορές υψηλότερο από την, τα αντίστοιχα τότε στην Αλία θάλασσα. Τώρα για το άλλο ερώτημα που ετέθη. Δεν έχουμε σαφή απάντηση γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάμε ε, με τις πράξεις, ε, τις εκτελεστικές πράξεις του Ταμείου. Στην ε, θαλάσσια αλία υπάρχει το μέτρο της ε, αποζημίωσης ε, της ζημιάς που έχουν προκαλέσει τα αρπακτικά ε, πουλιά. δεν ξέρω αν αυτό θα συμπεριληφθεί, αλλά καταρχήν μπορώ να πω ότι δεν καλύπτεται το άρθρο 42 αυτό το μέτρο. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβουμε μια τέτοια αποζημίωση. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται όμως καταρχήν δεν δείχνει να εμπίπτει στο άρθρο 42. Ευχαριστώ. Ωραία, δίνω το λόγο τώρα ξανά στην κυρία Νιούμαν για να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των αποθεμάτων, δεν το συμπεριέλαβα στην παρουσίασή μου γιατί αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν στόχο να, να συλλέξουμε πληροφορίες από 28 κράτη-μέλη. Όμως η κατάσταση είναι συγκρίσιμη με τα θαλάσσια αποθέματα. Ορισμένα αποθέματα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ορισμένα σε, μόνο, σε κάποιες χώρες μόνο, ιδιαίτερα σε παλαιότερα κράτη-μέλη, πολλά, πολλές περιοχές ε, έχουν φτωχύνει πολύ σε αποθέματα ε, ή δεν, ε, δεν διαθέτουν πλέον κανένα απόθεμα. Ήδη γίνονται προσπάθειες επαν... να εισαγωγής ε, συγκεκριμένων αποθεμάτων σε κάποιες περιοχές, οπότε πραγματικά δεν μπορώ να σας δώσω γενικά συμπεράσματα. Αυτό έχει σχέση και με τα αρπακτικά ζώα και ε, πουλιά. Ε, είναι σημαντική και η υπόλοιπη κοινωτική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ε, για αυτή για τα ε, ύδατα, η ΚΑΠ. Είναι οδηγίες οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη των ειδών στο υδάτινο περιβάλλον. Οπότε όταν βελτιώσουμε το υδάτινο περιβάλλον με άλλα μέτρα, τότε είναι πιο εύκολο να δούμε ε, πώς μπορεί να μειωθούν οι απώλειες μιας προκύπτουν από αυτά τα είδη, πουλιά και άλλα. Δηλαδή, ε, πώς είναι δυνατόν ε, να ρίχνουμε την ευθύνη σε άλλα είδη όταν εμείς δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χελιών. Η απαγόρευση ισχύει από το 2009. Οπότε παλιότερα γινόντουσαν εξαγωγές στην Ασία. Αλλά απαγορεύτηκαν. Ξέρω ότι γίνονται εξαγωγές και η παράνομη αλία είναι θέμα ε, για την ε, ε αλία. σίγουρα στην Πορτογαλία, αλλά ίσως και στον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Οκ, okay, ευχαριστούμε την κυρία Νιούμαν. Περνάμε στο σημείο 9 τη ημερησίας διάταξη. Παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β του ενημερωτικού σημειώματο με θέμα η κοινή αλληλευτική πολιτική διαδικασία επί παραβάση και επιβαλλόμενε κυρώσει στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε αυτό το σημείωμα, ανατέθηκε στην Blomeyer και Sands ε, και είναι εδώ παρόν σήμερα για να μας παρουσιάσει το σημείωμα. Ε, ο εκπρόσωπος της Blomeyer και Sands Έχετε το έγγραφο, το σημείωμα αυτό. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μάικ Μπέκε που θα μας το παρουσιάσει. 20 λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στην και Chance. Ε, Διεξαγάμε αυτή την ε, μελέτη για τις διαδικασίες επιπαραβάση και τις επιβαλλοντικές κυρώσεις. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν τους στόχους μας, μερικές πληροφορίες για την ε, κοινή ελευτική πολιτική και τις ε, διαδικασίες επιπαραβάση και τις ποινές, τα πορίσματά μας και κάποιες συστάσεις. Χωρίσαμε την έρευνα μας σε τρία κεφάλαια. Ε, καταρχήν μια ανασκόπηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους λειτουργούν οι διαδικασίες παραβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μηχανισμούς κυρώσεων, επιβολής κυρώσεων. Ξετάσαμε παραδείγματα των μελών. Και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε διαφορές σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να ε, προωθήσουμε την ισονομία και την ισοτιμία στον ανταγωνισμό. Καθώς επίσης και τον εναρμονισμό των, εναρμονισμό των κυρώσεων που εφαρμόζονται ε, στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για παράβαση των κανόνων της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Καταρχήν εξετάσαμε πότε εντοπίζεται η παράβαση και πότε ξεκινούν οι διαδικασίες επί παραβάση. Επίσης, εξετάσαμε και την φάση της επιθεώρησης του ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τις ε, επιθεωρήσεις, ε, ε, χρησιμοποιούνται συστήματα εισόδων-εξόδων, τεχνικά μέτρα. Επίσης διαπιστώσαμε ότι τα διάφορα κράτη-μέλη διαθέτουν ε, πολλές και διαφορετικές αρχές και σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα το Υπουργείο Αλληλείας, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων για θέματα εφαρμογής του νόμου, ε, Κάποιες άλλες φορές το Υπουργείο Άμυνας ε, όταν εμπλέκεται και το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό στις επιθεωρήσεις στη θάλασσα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε διάφορες αρχές που συμπράττουν. Έχουμε διαφορές μεταξύ των εθνικών ελεκτικών συστημάτων και το πώς λειτουργούν και δρούν οι διάφορες αρχ... αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ε, ε, μια πραγματικότητα που δημιουργεί και γραφειοκρατία αλλά και διακρίσεις. Απ' την άλλη μεριά περιπλέκει και την διαδικασία της προσπάθειας επιθεώρησης ε, και ελέγχου, δεδομένου ότι οι αρχές θα πρέπει να ε, επικοινωνούν μεταξύ τους κλπ. Οι κοινέ δράσεις ελέγχου που συντονίζονται από την κοινή υπηρεσία ελέγχου της Αλίας, κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της Αλίας, ε, αποτελούν την πλειοψηφία των ε, ευρωπαϊκών και εθνικών προσπαθειών. Οι, οι ε, έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην στεριά και όχι στη θάλασσα, ενδεχομένως για λόγους κόστους. Από την άλλη μεριά, στις επιθεωρήσεις που γίνονται στη θάλασσα εντοπίζονται περισσότερες παραβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της μας δείχνει με τα στοιχεία της ότι η πλειοψηφία των ε, παραβάσεων που εντοπίζονται στη θάλασσα σχετίζονται με αλλιευτικά εργαλεία, ενώ οι επιθεωρήσεις, οι επιθεωρήσεις έχουν σχέση και εντοπίζουν περισσότερο λανθασμένη ε, αναφορά στοιχείων, δεδομένων. Συμπεράναμε ότι και ο όγκος ε, των επιθεωρήσεων και η ποιότητα ε, επηρεάζουν τις κυρώσεις. Παρόλο ότι οι επιθεωρήσεις δεν εμπίπτουν στην στο πεδίο εφαρμογή, ε, στο, στο αντικείμενο τη έκθεση, θεωρούμε ότι οι επιθεωρήσεις έχουν άμεση σχέση με την ε, επιβολή κυρώσεων ε, και με την αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων. Έχουμε διάφορους τύπους παραβάσεων. Για παράδειγμα, σχετικές με αλληλευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ε, με κακή αναφορά των δεδομένων, ελλειπή δεδομένα. Μόλις εντοπίζεται κάποια ε, παράβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, αυτές μπορεί να είναι χρηματικά πρόστιμα. Υπάρχει και ένα point system, ε, όπου ε, όταν ένας αλίας συμπληρώσει το ανώτατο όριο πόντων, ε, το αφαιρείται προσωρινά η μόνιμα η άδεια. Και μάλιστα πολλές φορές, ε, μερικές φορές μάλλον, ε, μπορεί να επιβληθεί και ποινή φυλάκισης από δικαστήριο. Μεταξύ των πορισμάτων μπορούμε να πούμε και το εξή. Εξετάσαμε τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε ε, για την παρακολούθηση της ε, διαδικασίας παραβάση αφού εντοπιστεί η παράβαση. Δηλαδή η αρχή η οποία κάνει τι επιθεωρήσεις εντοπίζει μια παράβαση, ενημερώνει τι ε, αρμόδιες αρχές και αυτές οι αρμόδιες αρχές θέλουμε να δούμε τι κάνουν. αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, να δοθεί δηλαδή κάποια συνέχεια στον εντοπισμό παραβάσεων, στις στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι διοικητικές και όχι δικαστικές οι αρχές οι οποίες ε, επιβάλλουν τις ε, κυρώσεις. Αυτό έχει πολλές φορές ε, σχέση με τις διάφορες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών σε περιπτώσει σημαντικών παραβάσεων, ορισμένα έχουν και ποινικέ κυρώσει, προβλέπουν και ποινικέ κυρώσει. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερε ένομε τάξει προβλέπουν διοικητικέ κυρώσει από διοικητικέ αρχέ. Αυτό σημαίνει ότι οι ποινέ τι περισσότερε φορέ επιβάλλονται εξοδικαστικά. Οι διοικητικέ ε, κυρώσεις είναι ίσως ε, πιο οικονομικές. Ε, παρόλα αυτά, ενδεχομένως ε, είναι λίγο πιο επισφαλής με την έννοια ότι δεν, υπάρχει κάποιο, δεν εμπλέκεται κάποιο δικαστήριο. ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν διοικητικέ ε, ποινέ με βελτιωμένα συστήματα όμω. Αν δούμε τις εκτελεστικές αρχές, την, την αρχή η οποία επιβάλλει την ποινή, την αποφασίζει και την επιβάλλει, είναι συνήθως το Υπουργείο Αλληλεία. Ο Γενικός Γραμματέας, ε, Διευθυντής της ε, Αλληλευτική Διοίκησης, του Αλληλευτικού Τμήματος κλπ. Όμως κάποιε χώρε επιτρέπουν και σε αστυνομικέ αρχέ ή σε ε, σώματα επιθεωρητών ή λιμενικών να επιβάλλουν ε, οι ίδιοι τις ποινές. Η αρμοδιότητα για την ε, απόφαση διοικητικών κοινών, ε, διοικητικών ποινών μοιράζεται ανάμεσα σε διάφορες αρχές ή ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για τις ομοσπονδιακές δομής χώρες. Έχουμε διάφορους τύπους διοικητικών κυρώσεων. Ορισμένες κοινώσεις είναι ε, άμεσα εφαρμόσιμες και άλλες ε, κυρώσεις οι οποίες είναι συνοδευτικές. Οι άμεσα εκτελεστές κυρώσεις έχουν σκοπό να σταματήσουν αμέσως τη συνέχιση της παράβασης. και να κλείσει έτσι ο φάκελος. Οι πιο κοινέ διοικητικέ κυρώσει είναι τα πρόστιμα, χρηματικέ ποινέ, καθώ επίση και η αναστολή ή προσωρινή αναστολή τη αληπτική άδεια. Είναι παραδείγματα ε, ποινών που μπορούν αργότερα να επιβληθούν από διοικητικέ αρχές. Άλλε κυρώσει ε, μπορεί να είναι συνοδευτικέ μιας άλλης ποινική κύρωση, όπως για παράδειγμα η φυλάκιση, η οποία επιβάλλεται από δικαστήριο προφανώ. Αρκετέ χώρε έχουν και εναλλακτικά συστήματα επιλύση των διαφορών, για παράδειγμα εξοδικαστικά συστήματα, αλλά και την έκδοση προειδοποίησεων. Οι προειδοποιήσεις αποτελούν διακριτική ευχέρεια, βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια των επιθεωρητών, αλλά δεν είναι σαφείς οι όροι που χρησιμοποιούν, οι προϋποθέσεις οι οποίες δηλαδή εφαρμόζονται προκειμένου να εκδοθεί μια τέτοιου είδου προειδοποίηση από τις ε, διοικητικέ αρχές των κρατών μελών. Δεν διαφωνούμε με την χρήση της διακριτικής ευχέρειας γιατί οι επιθεωρητές είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις περιπτώσεις αυτές και μπορούν να αξιολογήσουν την περίπτωση, την κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το πότε και το πώ εκδίδονται τέτοιου είδου προειδοποίησεις, γιατί αλλιώς υπάρχει περίπτωση να γίνει κατάχρηση του συστήματος. Επίσης υπάρχει και το point system όπως σας είπα. Το σύστημα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει στις αρχές του 2012 τα κράτη-μέλη. Η δική μας έρευνα απέδειξε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο το point system. Ορισμένοι τύποι παραβάσεων παίρνουν συγκεκριμένο αριθμό πόντων και όταν συμπληρωθεί ένα μέγιστο ε, επιβάλλεται η, μια ποινή, μια κύρωση όπως η προσωρινή οριστική ε, αφαίρεση της άδεια. Το σύστημα αυτό θεωρείται καλό, θετικό, χρήσιμο τέτοιου είδου ε, ποινέ αντιμετωπίζονται θετικά αντίθετα με τις χρηματικές ποινές τις οποίες ο κλάδος θεωρεί ότι αυξάνουν το κόστος της αλίας. Επίσης ε, το point system δίδει τη δυνατότητα της άμεσης εφαρμογής της κύρωσης, ε, τα αποτελέσματά της φαίνονται αμέσως δηλαδή. Η εφαρμογή του point system όμως δεν γίνεται με μεγάλη διαφάνεια αυτή τη στιγμή. Δύσκολα εντοπίζει κανείς τις χώρες οι οποίες το εφαρμόζουν. Ορισμένες το έχουν εφαρμόσει και μας έδωσαν και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής του για κάποια μέτρα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Συνολικά όμως η εφαρμογή δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Παρόλο ότι μπορεί το μέτρο αυτό να έχει, το σύστημα αυτό να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Η χρήση των εξοδικαστικών συστημάτων επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το οποίο, παράδειγμα, οι αρχές προτείνουν στον κατηγορούμενο ε, να ε, συμβιβαστεί με μια χρηματική ποινή. Συνήθως ε, ή ο εισαγγελέας ή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, αλλά μερικές φορές υπάρχουν και συμβουλευτικές επιτροπές που το αναλαμβάνουν. Σε ορισμένε περιπτώσει τέτοιου είδου εξοδικαστική ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο για συγκεκριμένε παραβάσει και ε, για ε, την πρώτη φορά που κάποιο άτομο υποπίπτει σε συγκεκριμένη παράγραφαση. Είναι ένας τρόπος για να απελευθερωθούν τα δικαστήρια και μπορεί να είναι πράγματι χρήσιμο. Οι αρχές πολλές φορές χρησιμοποιούν την εξοδικαστική ρύθμιση για ε, συγκεκριμένο αριθμό παραβάσεων, όμως και εδώ υπάρχουν, υπάρχει κάποια διαφάνεια για το πώς χρησιμοποιείται, χρησιμοποιούνται τέτοιου είδου μέθοδοι. Δεν έχουμε στοιχεία ακριβή. Είναι ενισχυτικό αυτό. Είναι δύσκολο να εντοπίσουμε στατιστικά για το πόσο χρησιμοποιείται ένα τέτοιο εξοδικαστικό σύστημα από κάθε κράτος μέλος. Ένα πλεονέκτημα είναι οι επιπτώσεις, οι συνέπειες ε, για τους ε, παραβαίνοντες ε, τους κανόνες, ε, διότι η, μια δικαστική επίλυση θα καθυστερούσε πάρα πολύ ενδεχομένως. Σε ό,τι αφορά του διάφορου διάφορους κανόνες λειτουργίας, ορισμένα κρατημέλη χρησιμοποιούν αποκλειστικά ε, ποινικέ διαδικασίες, αλλά τα περισσότερα κρατημέλη διοικητικέ. Είναι σημαντικό όμως οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται να λαμβάνεται επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Επίσης είναι σημαντική η δυνατότητα έφεσης ή αναθεώρησης που θα επέτρεπε είτε, την ίδια, είτε η ίδια διοικητική αρχή είτε κάποια άλλη εξωτερική αρχή ή δικαστήριο να ξαναδεί την υπόθεση. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη του θέματος του, ε, των ένδικων μέσων που διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Ε, ορισμένες ε, νομοθεσίες έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, άλλες νομοθεσίες έχουν γενικές διοικητικές διαδικασίες που δεν έχουν σχέση μόνο με την αλία. Το σημαντικό όμως είναι να υπάρχουν διαδικασίες που να περιορίζουν ε, τη διακριτική ευχαίρεια των διοικητικών αρχών. Εξετάσαμε επίσης το, τη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάση. Και εδώ έχουμε σημαντική διακύμανση, διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. δεδομένου ότι ε, βιαζόμασταν δεν είχαμε χρόνο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αλλά βλέπουμε μεγάλη διάρκεια σε περιπτώσεις ποινικών διαδικασιών ενώ μικρότερη διάρκεια σε περιπτώσεις και συστήματα διοικητικών ποινών και κυρώσεων. Πάντως είναι σαφές ότι η μικρότερη διάρκεια αυξάνει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Διότι το αποτέλεσμα της κύρωσης γίνεται αμέσως αισθητό από τον παραβάτη. Τέλος έχουμε ένα κατάλογο συστάσεων. 22 συνολικά συστάσεων. 10 από αυτές τις βλέπετε εδώ. Είναι οι πιο σημαντικές. Πρώτον, βελτίωση συνεργασία μέσω τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου τη Αλία. Ε, βελτίωση συνεργασία ανάμεσα στι αρχέ επιβολή κυρώσεων και επιθεωρητών. Ένα τρόπο είναι μέσω τη υπηρεσία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Τσαλίας. Αυτή η σύσταση βασίζεται στο γεγονό ότι πολλοί επιθεωρητέ ανέφεραν πω δεν έχουν πλήρη εικόνα τι γίνεται μετά, μετά τον εντοπισμό της ε, παράβασης. Ε, δεν ξέρουν τι γίνεται από τα άλλα όργανα που επιφορτίζονται μετά. Τρίτον, βελτίωση της ε, συνεργασίας μεταξύ των ελεκτικών αρχών και των αρχών επιβολής κυρώσεων σε εθνικό επίπεδο. Και θα πρέπει να μοιράζονται και την ευθύνη της παρακολούθησης. Η Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, αλλά ε, θα πρέπει να τα δούμε μαζί. Θα πρέπει αυτά τα δύο επίπεδα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Τρίτη σύσταση να εξασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα για την παρακολούθηση των παραβάσεων. Θα πρέπει να δείτε συνέχεια σε όλες τις παραβάσεις, έτσι ώστε να μειωθεί η ατιμορρησία. Ε, η έλλειψη τέτοια παρακολούθηση υποσκάπτει την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος και ενδεχομένω δημιουργεί και ε, αρνητικές... Ε, αρνητική εικόνα του συστήματος στο κοινό. Τέταρτον, αποτελεσματικό σύστημα για την επιβολή κυρώσεων. Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα θα πρέπει οι κυρώσεις ε, να είναι αποτρεπτικές. Γιατί αλλιώς ε, μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Όπως σας είπα, για παράδειγμα, χρηματικές ποινές ε, εντάσσονται στον προπολογισμό της κάθε εταιρείας, δεν, επηρεάζουν την πρακτική πρόθεση της συμμετοχής άλλων κρατών μελών στις ελέγχους επιθεωρήσεις. Αυτό το μέτρο ε, μέσω του άρθρου 103.3 του εφαρμοστικού ανοισμού της ε, Κομισιόν δείχνει ότι η συμμετοχή αξιωματούχων άλλων κρατών μελών στους ελέγχους ε, είναι θετική ε, για τον κλάδο. Επίσης, ένα, ανάπτυξη ενός κοινού χρονοδιαγράμματος ε, κυρώσεων. Αυτό θα μπορούσε να συμφωνηθεί από τις εκτελεστικές αρχές των κρατών μελών και θα έδινε κάποιες κατευθύνες γραμμές στις αρχές ε, όταν πρόκειται για την ίδια παράβαση, έτσι ώστε να μην εξαρτάται από τον ίδιο τον εισαγγελέα, ας πούμε, ή την ε, κάθε διοικητική αρχή το τι ποινή θα επιβληθεί. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις διαδικασίες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το ποιοι κανόνες ακολουθούν σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων. Αυτό θα βελτίωνε την αμοιβία σύνδρομη μεταξύ των κρατών μελών και θα αύξανε την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων. Να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις στην επιβολή κυρώσεων. Θα πρέπει οι ποινές να επιβάλλονται έγκαιρα. 9. Ανταλλαγή πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται ως κυρώσεις. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το ποια μέτρα είναι διαθέσιμα και ποια κριτήρια και ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για την λήψη κάθε μέτρου. Αυτό για να αποφύγουμε ε, διαφθορά και παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων. Αυτά, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φράγα, κυρία Λεβίν, ο κύριος Ρωμέβα. Κυρία Φράγα. Ευχαριστώ πολύ του υπεύθυνου για αυτή την παρουσίαση, καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Είναι δύσκολο να λάβει κανεί ακριβείς πληροφορίε από τα κράτη-μέλη, γιατί τα θέματα αυτά είναι ευαίσθητα. Εργάστηκαν με τα στοιχεία που είχαν βέβαια. Οπότε η μελέτη είναι προφανώς περιορισμένη, δεν είναι δική του ευθύνη, οφείλεται στην πραγματικότητα. Εγώ θέλω να σχολιάσω το point system. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό ε, δεν τέθη σε εφαρμογή όταν έπρεπε. Κάποια κράτη-μέλη καθυστέρησαν πολύ, ενώ μερικά δεν ξέρουμε καν αν το έχουν εφαρμόσει και πώς το εφαρμόζουν. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας εξηγούσε που βρίσκεται το θέμα αυτό, τι κάνει για να παρακολουθήσει την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης από τα κράτη-μέλη. Γιατί εγώ επικρίνω πολύ τον κανονισμό ελέγχου, αλλά είναι κανονισμός, δεν είναι δυνατόν ένα τμήμα του να μην εφαρμόζεται ή να εφαρμόζεται καθυστερημένα. Το ερώτημα λοιπόν αφορά την Κομισιόν. Είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Δεν ήξερα ότι υφίσταται τέτοια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ήταν από τα πιο σημαντικά ε, σημεία της έκθεσης αυτής. Δεύτερον, τα ποινικά και διοικητικά συστήματα. Το διοικητικό σύστημα έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το ποινικό δικαστικό σύστημα, οπότε ενδεχομένως θα έπρεπε να γενικευτούν. Τώρα βέβαια αυτό είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Πρόκειται για συστάσεις. Όμως από την ανάλυση σας προκύπτει πως ε, υπάρχουν στοιχεία υπέρ του διοικητικού συστήματος το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια κλπ. κλπ. Όμως η ερώτησή μου, η βασική μου ερώτηση αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το point system. Δεδομένου ότι η μελέτη δείχνει πως το σύστημα αυτό είτε δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται μ, καθυστερημένα ή ελλειπώς. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Λεβίν. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε τις διαφορές ανάμεσα στο πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις ε, στην Αλία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και η κυρία Φράγα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στην εφαρμογή του συστήματος μορίων. Κάτι άλλο που ήθελα να ακούσω, αλλά μάλλον είναι δύσκολο να βρεθεί, θα ήταν μια σύγκριση ανάμεσα στις διάφορες παραβάσεις σύμφωνα με το σύστημα μορίων. Δηλαδή, στα διάφορα κράτη-μέλη ποιες παραβάσεις οδήγησαν ε, στο, στη συγκέντρωση των μορίων. Δηλαδή, αν ε, κάποιος ε, δεν αναφέρει τα αλλιεύματα, τι θα γίνει στη Φιλανδία, τι θα γίνει στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν ήταν δύσκολο για σας να βρείτε τα στοιχεία αυτά. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εάν θέλουμε να έχουμε δηλαδή ένα ενιαίο σχέδιο κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δούμε τη διαφορά στην εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη. Και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι σε κάποια κράτη-μέλη η κράτηση, η φυλάκιση αποτελεί επιλογή, νομίζω μέχρι τρία χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις. Φαίνονται, φαίνεται λοιπόν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, στην εφαρμογή. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω πώς τιμωρείται το ίδιο έγκλημα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και επίσης, όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων στην αλληλεία, η κυρώσεις δεν επιτρέπεται να είναι τόσο χαμηλές ώστε απλά να θεωρούνται κόστος λειτουργίας. Ε, δηλαδή, εάν το αλίευμα αξίζει ένα εκατομμύριο ευρώ και το πρόστιμο είναι 100.000 ευρώ, τότε ανά πάσα στιγμή θα προτιμούσε κανείς να το, να το διακινδυνεύσει. Ποιος είναι ο κίνδυνος, απλά να χάσει μέρος του κέρδους του. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρομέβα, ευχαριστώ πολύ. Όταν ε, στην προηγούμενη θητεία συζητήσαμε τον ε, κανονισμό περί ελέγχου, ένας από τους βασικούς μας ε, στόχους ήταν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ώστε η συμμόρφωση να αποτελεί βασική αρχή από μόνη της. Προφανώς γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ε, τελική ευθύνη. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή καθ' αυτή. Είναι κάτι που εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη, αλλά ε, τα προειδοποιήσαμε και το επιβεβαίνεται αυτό με τη, μελέτη, με τη μελέτη σας ότι υπάρχουν βασικές δυσκολίες σε αυτό. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον ε, τα κράτη-μέλη να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλα κράτη-μέλη μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν η δημιουργία των δικτύων αυτών μεταξύ των κρατών μελών. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, κάποια κράτη-μέλη ισχυρίστηκαν ότι μερικές φορές είναι θέμα διακριτικότητας. Να μην δίνει κανείς υπερβολικές πληροφορίες στους ανταγωνιστές. Αλλά μία είναι η ερώτησή μου. Αναφερθήκατε επανειλημμένα στον οργανισμό ελέγχου που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και τις κοινοποιεί. Εσείς πώς βλέπετε το παρόν επίπεδο του οργανισμού αυτού όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το προσωπικό. Ποιες είναι οι προοπτικές με αυτά που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, με εξέπληξε κάπως ότι στον κατάλογο χωρών που αναφέρατε για την επιβολή των κυρώσεων, δεν ξέρω αν δεν έχετε στοιχεία, ποιος είναι ο λόγος, δεν βλέπω την Ισπανία. Η ερώτησή μου είναι, αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν ε, οι σχετικές πληροφορίες επειδή δεν αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε την Ισπανία, επειδή είναι τόσο σήμαντα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Η Ισπανία είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά αλληλευτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήταν λοιπόν λογικό να συμπεριλαμβάνεται. Ερωτώ λοιπόν γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Γιατί τα κάνει όλα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να αναφερθεί ή και αυτή είναι η υποψία μου. Υπάρχει έλλειψη δεδομένων και συχνά έλλειψη πολιτικής βούλησης να παρασχεθούν τα δεδομένα. Θα παρακαλούσα λοιπόν να επιβεβαιώσετε αν η υποψία μου είναι σωστή ή όχι. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία του. Η μελέτη αυτή αναλύει αρκετά λεπτομερώς ε, το θέμα. Η Κομισιόν συμφωνεί συνολικά με τις συστάσεις περί ενίσχυσης ε, του συστήματος παρακολούθησης των κυρώσεων ενίσχυση των διαδικασιών και εφαρμογής αποτρεπτικών κυρώσεων στα κράτη-μέλη. Επίσης η μελέτη πολύ σωστά σημειώνει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τον, ε, προσδίδει τον θετικό ρόλο του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Επίσης θα συμφωνούσαμε με ένα σύστημα εναρμονισμένων αποτρεπτικών κυρώσεων. Αυτό θα βοηθούσε πολύ την αλία. Όμως, δεν έχουμε ολοκληρώσει τη λεπτομερή ανάλυση της μελέτης. Ξέρετε ότι η μελέτη αυτή έχει πολλές πληροφορίες και επηρεάζει όχι μόνο την Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Θεμάτων και Αλίας, αλλά και άλλες υπηρεσίες κομισιών. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση αυτή. σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει που έθεσαν οι ευρωβουλευτέ. Να σας δώσω κάποια στοιχεία παρόλο ότι δεν έχω συγκεκριμένη εντολή από τους ανωτέρους μου. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Φράγα καταρχήν. Για το point system. Η Καμισιόν η Κομισιόν αυτή τη στιγμή διενεργεί μια λεπτομερή ανάλυση του πώς εφαρμόζεται το σύστημα των κυρώσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Το point system αποτελεί τμήμα ενός πιο συνολικού συστήματος κυρώσεων. Και πολλές φορές το σύστημα των κυρώσεων ξεπερνάει τον τομέα της αλίας. Οπότε χρειάζεται να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε ποιος το έχει οθετήσει και ποιος όχι ή πώς, αλλά να δούμε και το πώς εφαρμόζεται και αν λειτουργεί. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Αφήσαμε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να κρίνουμε το αν εφαρμόζεται σωστά και αν δίνει αποτελέσματα. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη ερώτηση για την Κομισιόν. Απλά σχετικά με κάποια σχόλια που έγιναν. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Τσαλίας συνεργάζεται καθημερινά και στενά με τους εθνικούς επιθεωρητές. Μέσα στο πλαίσιο του κοινού προγραμματός επιθεωρήσεων που εφαρμόζει η Κομισιόν που ε, ε προγράμματα στα οποία ε, προβλέπεται η ε, συμμετοχή επιθεωρητών από άλλα κράτη-μέλη στους εθνικούς ελέγχους. Αυτή η συνεργασία λειτουργεί και δίνει καλά αποτελέσματα. Και μάλιστα η συνεργασία αυτή διευρύνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, επιθεωρήσεις από επιθεωρητές ενός κράτους μέλους γίνονται και σε ύδατα άλλου κράτους μέλους και μάλιστα σε σκάφη τα οποία δεν έχουν τη δική του σημαία. Οπότε βλέπετε ότι η συνεργασία αυτή διευρύνεται σταδιακά. Δεν νομίζω ότι απευθύνατε κάποια άλλη ερώτηση στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ξέχασα κάτι, πέστε μου το. Bien, muchas gracias. El eh, señor Rodus. Gea Rodust. Doch, ich meine, es ist gefragt worden und ich wiederhole das. Νομίζω ότι τέθηκε η ερώτηση και την επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Και υπόθηκε με μεγάλη σαφήνεια ότι στα διάφορα εθνικά κράτη επιβάλλονται διαφορετικές κυρώσεις. Σε κάποια κράτη-μέλη επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σε άλλες μπορεί να καταλήξω στη φυλακή ως αλίας. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Κομισιόν και νομίζω τέθηκε με σαφήνεια η ερώτηση είναι η Κομισιόν το γνωρίζει αυτό και πώς χειρίζεται το θέμα. Θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και ο Αλίας στο κάτω-κάτω τι θα κάνει. Δηλαδή εγώ αν είμαι ψαράς να αλλιεύω μόνο σε ένα κράτος μέλος όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και όπου δεν κινδυνεύω να καταλήξω στη φυλακή. Ε, βρίσκω ότι είναι πολύ δύσκολο το θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ που το ε, περιγράψατε με τόση σαφήνεια. Η μάλιστα πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό εν μέρει έχει ήδη απαντηθεί από τη μελέτη. Η αρμοδιότητα αυτή ε, βαραίνει τα κράτη-μέλη η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την ε, δημιουργία ενός κοινού συστήματος, για την θέσπιση ενός κοινού συστήματος που θα περιλαμβάνει κοινέ πρακτικές από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε οι κυρώσεις να είναι ισοδύναμου αποτελέσματος και επίσης να είναι επαρκώς αποτρεπτικές. Παρ' όλα αυτά, οι κυρώσεις αποτελούν δικαιοδοσία των κρατών μελών. Έχουμε εργαστεί ε, προς την κατεύθυνση ενός κοινού συστήματος, αλλά χωρίς πολλά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Μπέκε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Το point system που αναφέρατε αρκετές φορές έχει μεγάλο δυναμικό κατά τη γνώμη μου και η εφαρμογή του συστήματος δεν κινείται με τους ίδιους ρυθμούς στα διάφορα κράτη-μέλη. Όπως είπε και η Κομισιόν, ας του δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά είναι σημαντικό γιατί η ιδέα πίσω από το point system είναι να έχουμε παρόμοιες κυρώσεις για την ίδια παράβαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα επιληθεί το πρόβλημα που ανέφερε η προηγούμενη Ευρωβουλευτής. Θα αποφύγει τη μετανάστευση των παραβατών από τη μία περιοχή στην άλλη λόγω των διαφορετικών κυρώσεων. Γιατί αν έχεις το ίδιο πρόστιμο ή την ίδια ποινή στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μεσόγειο, δεν υπάρχει λόγος να έχεις τέτοια οπορτουνιστική συμπεριφορά, να να φεύγεις για να αποφεύγεις τις πιο αυστηρές τιμωρίες. Το βασικό θέμα είναι η αρμοδιότητα που την έχει το κράτος μέλος για την υποβολή των κυρώσεων. Οι συστάσεις εστιάζουν στη βελτίωση της εναρμόνισης μέσω των μέτρων ε, κυρώσεων. Οι εισαγγελείς έχουν μία βάση δεδομένων για προηγούμενες ε, ποινές που επιβλήθηκαν σε αλληλείς, ούτως ώστε να μην έχουμε υποτροπίαση από μέρους τους και ούτως ώστε να έχουμε αντίστοιχες κυρώσεις και στο μέλλον επίσης. Επίσης, η σημασία της κοινοποίησης των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα μας επιτρέψει τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, τη διαβίβαση σε ένα άλλο κράτο σημαία, Φερρυπίν, και την εξασφάλιση ότι δίδονται επαρκείς πληροφορίες, ούτως ώστε να τιμωρηθεί παράβαση και στην άλλη χώρα. Ακούσαμε παραδείγματα όπου οι εκθέσεις των επιθεών δεν έγιναν αποδεκτές δεν θεωρήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τον εισαγγελέα, λόγω του ότι προέρχονταν από άλλη χώρα. Αυτά τα στοιχεία τα αντιμετωπίζει η κοινή αλληλευτική πολιτική. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος επ' αυτών. Το να υπάρξει αυτή η συνειδητοποίηση μεταξύ των αρχών ότι χρειάζονται κάποιες πληροφορίε ούτως ώστε να δίδουν τις πληροφορίε που χρειάζονται για να αποφύγουν τα προβλήματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επίπεδο των κυρώσεων τώρα. Πολύ σημαντικό θέμα, προφανώς. Μακάρι να είχαμε περισσότερες ε, πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη. Μερικά από τα παραδείγματα που σας έδωσα προέρχονται από δεδομένα που μαζέψαμε μέσα από το δικό μας desk research και μέσα από έρευνες που κάναμε. Παραδείγματο χάρη ε, στο Βέλγιο. Ε, σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο Φλάνδρα, οι ευρωβουλευτέ ζήτησαν, οι βουλευτέ οι Βέλγοι, συγγνώμη, ζήτησαν αυτέ τι προφορίε από του υπουργού. Και οι υπουργοί απάντησαν ότι είναι δύσκολο να κάνουμε μια κατανομή, να δούμε ποια ποινή παίρνει επισύρει τέτοια κύρωση. Έχουμε το συνολικό ποσό, αλλά όχι το επιμέρους ποσό. Επίσης, η κοινοβουλευτική ε, επιτήρηση και έλεγχος είναι πολύ σημαντικό. Σε εθνικό επίπεδο το, η Βουλή, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα όπως έκαναν ας πούμε οι φλαμανδοί ε, βουλευτές στον Υπουργό. Πόσες παραβάσεις υπήρξαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Ένα άλλο θέμα σε επίπεδο κυρώσεων το οποίο το έχουμε συζητήσει, είναι ότι όταν ε, κάποιος κερδίζει περισσότερο από την παράβαση παρά από την καταβολή του προστίμου, προφανώς εθαρρύνεται η παραβατική συμπεριφορά. Μπορούμε να έχουμε βέβαια μια στάση που να βασίζεται περισσότερο σε μια ηθική συμπεριφορά ε, αλλά αυτό βασίζεται περισσότερο στην αυτορύθμιση του κλάδου. Είναι ένα άλλο θέμα. Είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο εδώ. Με βάση τα πορίσματά, βάση τα πορίσματά μας, καλό είναι να υπάρχει και η αυτορύθμιση. Δηλαδή, επιμερισμός των πόρων, θερυπίν, ε, είναι ένα πράγμα που μπορεί να λειτουργήσει καλά. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην αυτορύθμιση για να βελτιώσουμε την ε, συμμόρφωση και η οριοθέτηση λοιπόν ανάμεσα σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο της επιβολή των κυρώσεων δεν είναι τόσο σαφή. Τα στοιχεία για την Ισπανία τα ζητήσαμε. Και είχαμε δώσει και προθεσμία μέχρι τέλος, μάλλον από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Δεκεμβρίου. Δεν ήταν μεγάλη περίοδος όταν συλλέγουμε γενικά δεδομένα για τις καταδίκες, για διάφορα είδη παραβάσεων και ποινικών αδικημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι δύσκολο. Ε, είναι δύσκολο να έχουμε τα συνολικά στοιχεία. Ε, Παραδείγματο χάρη στην Ισπανία, για τι περιπτώσει διαφθορά, α πούμε. Συγκεκριμένα δεδομένα για τι καταδίκε, σε αυτά δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Αν δούμε λοιπόν τώρα τις παραβάσεις στην Αλία, στην Ολλανδία ο δημόσιος κατήγορος για περιβαλλοντικά θέματα είναι ο αρμόδιος. Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τις, τον αριθμό των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, αλλά δεν ξέρουμε στην Αλία πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν στον τομέα της Αλίας. Καλό είναι να υπάρχουν λοιπόν καλές πληροφορίες για να καλυφθούν αυτά κενά σε όλα αυτά τα επίπεδα. Για τον, την υπηρεσία ελέγχου της αλίας και τι απήχηση έχει, τι αντίληψη υπάρχει για αυτή. Από την αξιολόγηση που της έγινε δείχνει ότι πρόκειται για μια ελεγκτική υπηρεσία των ελεγχτών. Έχει ένα πρόβλημα όμως πόρων. Ε, οι έρευνε είναι πάρα πολύ ακριβές όταν γίνονται στη θάλασσα, Φερρυπίν. Άκουσα ένα παράδειγμα εκτιμήσεων και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό το νούμερο, αλλά στην Ολλανδία, ας πούμε, μία μέρα επιθεώρηση κοστίζει 10.000 ευρώ. Πολλέ από αυτέ τι ε, επιθεωρητικές υπηρεσίες, ε, ελεγκτικέ υπηρεσίες, ας πούμε, ε, αντιμετωπίζουν αναδιάρθρωση. Ε, ε, στην Ολλανδία είχαμε μείωση των πόρων λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας και αυξημένη δραστηριότητα. Άρα υπάρχει μεγάλη πίωση. Δεν έχουμε κοιτάξει του πόρου τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου και να εκτιμήσουμε κατά πόσον είναι επαρκή η πόρη. Ε, επίσης, τι γίνεται με την αρμοδιότητα για επιβολή κυρώσεων ως κράτους μέλους. Ε, η υπηρεσία αυτή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιθεώρηση και στην, στις Δηλαδή, γίνεται η επιθεώρηση και μετά πώς θα φτάσουμε στην κύρωση. Ένα άλλο θέμα που αναφέρει η έκθεση, ενδεί παραδείγματος, ορισμένες από αυτές τις ελεγκτικές υπηρεσίες καλύπτουν περισσότερες πτυχές, όχι μόνο την αλληλεία, αλλά την ασφάλεια των τροφίμων, ε, τα κτηνιατρικά, ε, θέματα φυτών, διάφορες επιθεωρήσεις, διάφορες μορφές ε, επιθεωρήσεων σε διάφορους τομείς. Και οι οι επιθεωρητικές υπηρεσίες ασχολούνται και με τις εξαγωγές, φερειπίνη τι εξαγωγές. Το ερώτημα είναι, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Αυτή τη στιγμή ε, μία υπηρεσία επιθεώρησης κάνει οποιαδήποτε επιθεώρηση και επιστοπεί εν συνεχεία και τη βιομηχανία έναντι πληρωμής. Όχι για να βγάλει κέρδος, αλλά για να καλύψει κάποια έξοδα. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση των πόρων που έχουν αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να δημιουργήσει θέμα ακαιρεότητας και ανεξαρτησίας και σοβαρή και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων τη. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Όχι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Σταματούμε εδώ την συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα.